Dear colleagues, we have some delay, but I think that we can. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε λίγο καθυστερήσει. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις συνεδρίες της Επιτροπής μας. I'm not able to see the rapporteur. Αλλά δεν βλέπω τον Δεν Λοιπόν, το πρώτο θέμα στη μέση διάταξη είναι η μείωση των εθνικών ε, εκπομπών ορισμένων ε, ρηπαντών της ατμόσφαιρας. Είναι τμήμα της οδηγίας για καθαρό αέρα που ανήγγειλε η Κομισιόν το Δεκέμβριο του 2013. Θέμα λοιπόν που μας ε, έχει απασχολήσει ως ένβη και από την προηγούμενη θητεία, η τρίτη ανταλλαγή απόψεων έγινε στην Επιτροπή μας <clears throat> στις 19 Τρίτου 14 και κατόπιν οι συντονιστές αποφάσισαν να συνεχιστεί ως γραπτή διαδικασία η οποία κατέληξε πριν από τις εκλογές του Μαΐου. και ζήτησα να κάνει το Κοινοβούλιο μια συμπληρωματική μελέτη αντικτύπου για την συσχέτιση αυτού του μέτρου με το πλαίσιο για το κλίμα και το περιβάλλον 2030. Αυτή η μελέτη αντικτύπου εκπονήθηκε και έχουμε εδώ αντίγραφα. Οπότε περιμένουμε την εισηγήτρια, η οποία όμως δεν είναι ακόμη εδώ. I've seen uh, the rapporteur. Α, ειδού η εισηγήτρια. Τζούλη. και τις δίνω το λόγο και μετά θα μας μιλήσει και ο συντάκτης της συμπροματικής έκθεσης αντικτύπου. Τζούνι παρακαλώ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα πω πολλά σε αυτή τη φάση. Γιατί το σημαντικό θέμα που πρέπει να συζητήσουμε σήμερα είναι συμπληρωματική μελέτη αντικτύπου. Ελπίζω να την έχετε όλοι λάβει. Είναι αρκετά μεγάλο κείμενο. Όπως ξέρετε το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα τεχνικό και πριν ε, ως Επιτροπή αισθανθούμε σε θέση να καταλήξουμε σε μια συνενετική άποψη είναι πολύ σημαντικό οι συνάδελφοι να μπορέσουν να εξετάσουν, να κατανοήσουν τα τεχνικά στοιχεία. Διότι κατά τις συζητήσεις που έχω ήδη διεξάγει με τους κοιόδης, με τα κρατημέλη, όλα όσα πρέπει να κάνει κανείς ως εισηγητής, έχω καταλάβει σαφώς ότι η συζήτηση θα εστιάσει στο εάν και κατά πόσο είναι αποδεκτές οι στατιστικές που έχουμε, γιατί κάποια κράτη-μέλη θα τις αμφισβητήσουν. Αυτή τη στιγμή που το συζητάμε εδώ, κάπου σε κάποια υπηρεσία κάποιου κράτους μέλους ε, αμφισβητούνται αυτές οι στατιστικές. Η μελέτη αντικτύπου λοιπόν που ε, προετοίμασε η δική μας υπηρεσία θεωρώ ότι είναι η πιο αναλυτική εξάντε έκθεση που έχουμε λάβει ποτέ. Γι' αυτό ζήτησα πολύ συγκεκριμένα να συμπεριληφθεί αυτή η έκθεση στην ημερήσια διάταξη για να τη συζητήσουμε όλοι, να έχουμε λάβει όλοι τις ίδιες διευκρινήσεις για να την αξιοποιήσουμε ως βάση συζήτησης. Εάν λοιπόν συμφωνείτε, καλό θα ήταν να περάσουμε απευθείας από τους υπευθύνους της ε, έκθεσής τους και μετά βεβαίως ε, οι συνάδελφοι θα παρέμβουν. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Πριν ε, περάσουμε στην παρουσίαση, να καλωσορίσω πέντε τοπικά εκλεγμένους από την κάτω Σαξονία, που είναι παρόντες στη συνεδρίασή μας. Τους έχει προσκαλέσει η συνάδελφος Μάισνα και ο συνάδελφος... Α, η Μάισνα μόνο, μάλιστα. Γιατί είναι από την περιοχή της. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Να δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στον κύριο Μάρκους Αμάν. που συνέταξε αυτήν τη συντορματική έκθεση αντικτύπου για να μας εξηγήσει το αποτέλεσμα, τα αποτελέσματα της μελέτης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπατε, η υπηρεσία μου διεξήγαγε μια συμπληρωματική έκθεση αντικτύπου. Ασχολούμενη κυρίως στην αλληλεπίδραση μεταξύ της, ποιότητας, της πολιτικής της Ένωσης για την ποιότητα του αέρα και της πολιτικής της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια. Έχετε το γραπτό κείμενο. Είναι ιδιαίτερα αναλυτικό. Τώρα να συνοψίσω τα κύρια ευρήματα. Σε τι πλαίσιο διεξήχθη η έκθεση πολύ ισχυρή αλληλεπίδραση των ατμοσφαιρικών, των ατμοσφαιρικών ρήπων και των αερίων ε, θερμοκηπίου. Γιατί προκύπτουν από τις ίδιες πηγές. Ό,τι κάνει κανείς για τις πηγές, κυρίως την κατανάλωση ενέργειας ή για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίων, των ατμοσφαιρικών ρήπων, λοιπόν, θα έχει επιπτώσεις και παρενέργειες στις άλλες πλευρές. Αν μειώσουμε τα αέρια θερμοκηπίου, Πρέπει κάτι να κάνετε λοιπόν ε, για την παραγωγή ενέργειας, άρα μειώνετε τους ατμοσφαιρικούς ρήπους. Μα ζητήσατε κυρίως να εξετάσουμε τις επιπτώσεις των πρόσφατων ε, προτάσεων για την ποιότητα του αέρα σε σχέση με τις ακόμη πιο πρόσφατες αποφάσεις για τους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια. Ο όγκος και η δομή της χρήσης ενέργειας καθορίζουν δύο σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, το κόστος για τα επιπλέον μέτρα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, το οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις προτάσεις της Κομισιόν, αυτό το κόστος. Αυτό βεβαίως επηρεάζει και το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνονται τα περαιτέρω μέτρα. γιατί το περιθωριακό κόστος ε, σε σχέση με το περιφερειακό όφελος είναι το καθοριστικό για να λαμβάνονται αποφάσεις. Το 2013 η Επιτροπή πρότεινε την οδηγία NEC. Η ανάλυση και, το, και η μελέτη αντικτύπου βασίστηκε στο Primes 2013 που ήταν μια πρόβλεψη για την ενέργεια με βάση τα στοιχεία του 2012 και συμμετείχε τα στοιχεία της πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα της Ένωσης από το, την άνοιξη του 2012. Το 2014 η Επιτροπή πρότεινε νέους στόχους για την ενέργεια και το κλίμα. Αυτό επιβεβαιώθηκε πρόσφατα και από τα πορίσματα του Συμβουλίου. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό θέμα τώρα. Τι επιπτώσεις θα έχουν αυτοί οι νέοι στόχοι στο πακέτο για το καθαρό ατμοσφαιρικό αέρα, για την καθαρή ατμόσφαιρα. Έχουμε ξανακάνει τέτοια ανάλυση και χρησιμοποίησαμε το ίδιο μοντέλο, τις ίδιες δυνατότητες, τα ίδια στοιχεία με τη μελέτη για την ποιότητα του αέρα και αναλύσαμε τις διαφορές και επιπτώσεις των νέων λοιπόν αυτών στόχων την ενέργεια και την έρευνα. Χρησιμοποίησαμε λοιπόν ένα σενάριο που χρησιμοποιήθηκε και για την ανακοίνωση της Κομισιόν για το πλαίσιο πολιτικής κλίματος μέχρι το 2030. Είναι το GHG 40 κάθετος EE. E. Αυτό το σενάριο είναι πολύ κοντά στην πρόταση της Επιτροπής για τα αέρια θερμοκηπίου, δηλαδή μείον 40% το 2030. προτείνεται 26,4% για τα ανανεώσιμα, για τις ανανεώσιμες και 29,3% και 29 αποδοτικότητα της ενέργειας για το 2030. Αξιοποίησαμε λοιπόν αυτό το σενάριο, αλλά απλώς αλλάξαμε την πρόβλεψη για την ενέργεια με τα νέα στοιχεία που θα μας επέτρεπαν να επιτύχουμε τους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν ε, δούμε τώρα την κατανάλωση ενέργειας, το νέο σενάριο είναι οι νέοι στόχοι που θα είχαν ε, αποτέλεσμα ένα μείον 10% σε σχέση με την ε, προηγούμενη πρόβληψη για το 2030. Η πιο σημαντική μείωση προκύπτει λόγω του φυσικού αερίου και βελτιώσεις της αποδοτικότητας ιδίως στον τομέα των νοικοκυριών μέσω καλύτερης μόνωσης κτλ. Εδώ, σε αυτό το διάγραμμα, βλέπετε τις επιπτώσεις ιδίω το όφελος που θα προκύψει από τα επιπλέον μέτρα που προτείνει η Επιτροπή με βάση τους νέους στόχους. Είναι ένα διάγραμμα επιστημονικό που συνοψίζει τα κύρια στοιχεία τι έχουμε επιλέξει στους άξονες. Στον κάθε το άξονα βλέπετε την επίπτωση επί της υγείας το 2030 και όσο πηγαίνετε προς τα δεξιά έχουμε λιγότερους θανάτους, αυξάνεται το βιώσιμο αλλά βλέπετε πως αυξάνεται και το κόστος. Η διακεκομένη κόκκινη γραμμή δείχνει πόσο αυξάνεται το κόστος με την πρόταση της Επιτροπής με σημείο αναφοράς την πρόταση της Επιτροπής. Βλέπετε πώς ανεβαίνει λοιπόν το κόστος και μάλιστα πόσο πιο έντονα αυξάνεται το κόστος. Ενώ η συνεχής γραμμή δείχνει το συνολικό κόστος της ενέργειας της προτάσης Επιτροπής. Η μπλε γραμμή μάλλον το μπλε εμβαδόν, το γαλάζιο εμβαδόν, δείχνει τα ωφέλη επί της υγείας ε, από πλευράς οικονομικής. Βλέπετε λοιπόν ένα ολόκληρο πλαίσιο, ένα ολόκληρο εμβαδόν. Το ουσιώδες ποιο είναι. Ότι τα περισσότερα μέτρα θα μας δώσουν ε, ωφέλη επί της υγείας που κατά πολύ υπερβαίνουν το κόστος. Η συνεχής ε, μπλε γραμμή είναι η στόχη της Κομισιόν. Στόχος μας είναι το 60% των κομμέτρων. Τι είναι σημαντικό εδώ. Είναι η συνεχής κόκκινη γραμμή που δείχνει το κόστος του πακέτου κλίματος και ενέργειας. Αν έχουμε λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και λιγότερους ρηπαντές, βλέπουμε ότι το κόστος είναι χαμηλό, 3,5 δις ευρώ ανά έτος λιγότερο από ότι το κόστος με το προηγούμενο σενάριο, τελικά 22% της βελτίωσης επί της υγείας θα προκύψει αυτόματα ως παράπλευρο όφελος από την εφαρμογή των στόχων της ενέργειας και του κλίματος, χωρίς συμπληρωματικό κόστος. Θα έχουμε όφελος 3,5 δις το χρόνο. Αυτό είναι το νέο σημείο εκκίνησης για την επίτευξη των στόχων κλίματος ενέργειας και αν ε, μειώσουμε περισσότερο, αυξάνεται το κόστος. Μειώνουμε τους ε, ατμοσφαιρικούς ρυπαντές πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν δυνατόν με τις προηγούμενες προβλέψεις για την ενέργεια που δεν συμπεριλάμβαναν στόχους για την ενέργεια. Επίσης βλέπετε, η κάθετη γραμμή είναι το επίπεδο το φιλόδοξο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό σημαίνει ουσιοδός μικρότερο κόστος. Το σημείο αποκοπής μεταξύ, το σημείο μη δηλαδή, μεταξύ της συνεχούς κόκκινης γραμμής και της μπλε γραμμής είναι κάτω από το 0. Δηλαδή, το κόστος εφαρμογής αυτής της νέας πολιτικής είναι μικρότερο από το κόστος εφαρμογής της αρχικής πολιτικής. Για να δούμε εδώ στο επόμενο slide για να καταλάβουμε καλύτερα. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία. Εδώ έχουμε έναν απλό πίνακα. Εδώ έχουμε μια σύγκριση του κόστους στην, ε, στην αριστερή στήλη το νέο σενάριο, στη δεξιά στήλη το παλιό σενάριο. Το κόστος ε, της ε, εφαρμογής της τρέχουσας νομοθεσίας έως το 2030 είναι 90,2 στην περίπτωση αναφοράς μειώνεται και πηγαίνει στα 86,6 δις. Και μετά έχουμε και το επιπλέον κόστος για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους της Επιτροπής. Αυτό είναι 3,3 ενώ οι ίδιοι στόχοι, η ίδια βελτίωση της υγείας θα μπορούσε να επιτευχθεί με τους στόχους ενέργειας ε, κλίματος με συμπληρωματικό κόστος 1,4 δις. Άρα συνολικό κόστος από τη μία πλευρά 88 για το πακέτο κλίματος ενέργειας, ενώ είναι 93,5 στην περίπτωση αναφοράς. Άρα 5,5 δις λιγότερα. Σαφές πόρισμα. Οι νέοι στόχοι κλίματος ενέργειας βελτιώνουν την υγεία και μπορούν να επιτευχθούν με χαμηλότερο κόστος. Βλέπετε εδώ το κόστος είναι ακόμη χαμηλότερο, 88 δις. Χαμηλότερο κόστος από αυτό που δαπανούμε τώρα για να εφαρμόσουμε την τρέχουσα νομοθεσία που βασίζεται στο παλιό σενάριο για την ενέργεια. Αυτά για το κόστος, για να επιτύχουμε τους προτινόμενους στόχους. Επίσης, η Επιτροπή σας μας ζήτησε να κάνουμε μια οικονομική ανάλυση του οικονομικά βελτίστου επίπεδου θα ήταν, ποια θα ήταν μια λογική φιλοδοξία. Πώς γίνεται αυτό. Αυτό συμβαίνει όταν το περιθωριακό κόστος ισούται με το οικονομικό όφελος, με το, συγγνώμη, με το περιφερειακό όφελος. Εδώ βλέπετε το περιθωριακό κόστος σε σχέση με το περιφερειακό κέρδος ή όφελος. Η συνεχής γραμμή είναι η γραμμή του περιθωριακού κόστους για την επίτευξη των στόχων κλίματος ενέργειας και το μπλε εμβαδόν είναι το ενδεχόμενο ε, ωφελημάτων επί για την υγεία. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με την παλιά πρόταση, όχι την τρέχουσα πρόταση της Κομισιόν, 67% βέλτιστο επίπεδο, εκεί λοιπόν που το περιθωριακό κόστος και όφελος είναι το ίδιο, είναι στο 75% μείωση του χάσματος, ενώ η διακεκομένη γραμμή είναι το όριο για το μπλε εμβαδόν, είναι μεταξύ 75 και 92. Η πρόταση της Κομισιόν θέλει να μειωθεί το χάσμα μεταξύ 67, κατά 67% μέχρι το 2030. Είναι 5% κάτω από το βέλτιστο. Αυτό από ό,τι κατάλαβα ήταν αποτέλεσμα των ε, διαπραγματεύσεων. Αποδέχθηκε η Κομισιόν λοιπόν να υπάρξουν 5 έτη παραπάνω για να εφαρμοστεί ένα στόχος κατά 5% χαμηλότερος. Οπότε θέλουμε μείωση του χάσματος κατά 67%. Ενώ το βέλτιστο επίπεδο με βάση την παλιά πρόταση ήταν <coughs> μεταξύ 75 και 92. Για να δούμε τώρα την ε, συνεχή γραμμή που μας λέει ότι το νέο σενάριο μπορεί να πάει μέχρι και 106% σε σχέση με το αρχικό σενάριο. Αυτό είναι πολύ πιο φιλόδοξο από την πρόταση της Κομισιόν. για να δούμε ποια είναι η πιο συντηρητική τώρα αποτίμηση του ωφέλους. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτήν την πιο συντηρητική 92% και την πρόταση της Κομισιόν είναι περίπου, είναι περίπου 16 με χιλιάδες προώρων θανάτων ανά έτος. Άρα, εάν εφαρμόσουμε αυτές τις νέες προτάσεις, θα έχουμε 17.000 λιγότερους προώρους θανάτους. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία. Είπα λοιπόν ήδη, γιατί έχουμε διαφορετικούς τρόπους να εκφράσουμε το όφελος επί της υγείας. Θα μπορούσαμε να πούμε 140.000 ε, έτη ζωής ή αν θέλουμε να το εκφράσουμε σε αριθμό προώρων θανάτων, 16.200 περιπτώσεις λιγότερων. Ποιο είναι το συνολικό κόστος ατμοσφαιρικής ρήπανσης, θα ήταν 91,3 δισεκατομμύρια αντί για 93,5, δηλαδή 2,2 δισεκατομμύρια λιγότερο ανά έτος. Και το ωφέλη επί της υγείας, αν τα εκφράσουμε νομισματικά θα ήταν 8,4 ε, ε, έως 50,8 δισεκατομμύρια. Και τέλος καταλήγω. Βλέπουμε λοιπόν ότι με βάση το σενάριο κλίματος ενέργειας το κόστος ελέγχου της ρήπανσης για να επιτύχουμε τους στόχους υγείας της Κομισιόν θα ήταν 5,5 δισεκατομμύρια λιγότερο έναντι του παλαιού σενάριου και η βέλτιστη οικονομική κατανομή πόρων για τους ε, στόχους κλίματος ενέργειας θα μας προσέθεται 140.000 έτη ζωής και το συνολικό κόστος ε, ελέγχου της ατμοσφαιρικής λίπανσης θα ήταν κατά 2,2 δισεκατομμύρια λιγότερο με βάση ε, σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν και τα συμπληρωματικά ε, ωφέλη για την υγεία θα ήταν 8,5 έως και 50 δις περισσότερο. Για το 2020 η Κομισιόν δεν έχει κάνει πρόταση για ανώτατα όρια εκπομπών. Αλλά εάν προσπαθήσουμε να ε, κάνουμε μια πρόβλεψη με βάση ένα λογικά αισιόδοξο σενάριο, λογικά φιλόδοξο σενάριο, θα είχαμε ωφέλη μεγαλύτερα από το αναθεωρημένο πρωτόκολλο του Gothenburg, που θα πήγαιναν από 40 έως και 300 δις. Υπάρχουν πολύ περισσότερα στοιχεία στο έγγραφο που έχετε ενώπιόν σας και με χαρά να απαντήσω στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Αφού ακούσαμε λοιπόν αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη αντικτύπου, θα δώσω το λόγο στους και συζητητές των πολιτικών ομάδων κυρία Γκαρδίνη από το ΕΛΚ ε, μου ανέθεσε το ρόλο αυτό. Έτσι λοιπόν θα μου δώσω το λόγο και θα σας πω ποιες είναι οι αντιπώσεις μου. Καταρχήν ευχαριστώ τον Κινόμαν για αυτή τη μελέτη που αφενός μας αποσαφηνίζει ποιες είναι οι πολύ θετικές σχέσεις μεταξύ των δύο πολιτικών και αφετέρου μας δίνει και κάποια χρήσιμα στοιχεία αξιολόγηση. Φυσικά προκύπτει από ότι μεταξύ των δύο πολιτικών υπάρχουν θετικές συνέργειες, δηλαδή η εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής και των νέων προτάσεων για το κλίμα και την ενέργεια έχουν θετικό αποτέλεσμα, θετικό αντίκτυπο επί της πρότασης ε, της ε, πολιτικής σε ό,τι αφορά την ατμοσφαιρική ρήπανση και την ποιότητα του αέρα. Έχουμε θετικά αποτελέσματα και σε ό,τι αφορά την υγεία και έχουμε και πολύ μεγάλη εξοικονόμηση. Δηλαδή, μιλήσατε για 140.000 έτη ζωή, πάνω από 7% σχέση με την πρόταση Κομισιόν. Μιλήσατε για τη μείωση του κόστου 2,3 ε, δισεκατομμύρια ευρώ. Και επίση, ε, ωφέλει 8,5 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον σε ό,τι αφορά τα ωφέλη για την υγεία. Και φυσικά είναι σαφές ότι για μας ως Επιτροπή είναι καλό να τα γνωρίζουμε αυτά τα πλεονεκτήματα και επίσης και για την αξιολόγηση που θα κάνουμε επί άλλων πολιτικών γιατί είναι φυσικά, φυσικό ότι αν υπάρχουν ωφέλη σε αυτή την πολιτική σημαίνει ότι θα υπάρχει μικρότερο κόστος και για την εφαρμογή άλλων πολιτικών. Πρέπει ακόμη να πω ότι οι θετικές συνέπειες ε, οθούν την ομάδα μας να κάνει θετική αξιολόγηση αυτής της μελέτης, αλλά πιστεύω βεβαίως ότι σε όλα τα μέλη της Επιτροπής μας θα μπορούσαν να δοθούν τα στοιχεία αξιολόγησης για αυτή τη δέσμη μέτρων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που θα κληθούμε να αξιολογήσουμε και να εγκρίνουμε για την ομάδα των σοσιαλιστών. Θα έδινα το λόγο στη συνάδελφο Ντάνς και κατόπιν θα συνεχίσουμε και με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά που κάνατε για την παρουσίαση αυτής της μελέτης αντικτύπου επιβεβαιώνοντας τα αμοιβαία ωφέλη που υπάρχουν, όταν συνδυάσουμε το πολιτικής, βλέπουμε ότι η μείωση του κόστους που μπορεί να επιτευχθεί σε συνδυασμό με τα ωφέλη για την υγεία είναι πραγματικά κάτι φανταστικό. Δηλαδή να μπορούμε να πούμε ότι αν έχουμε ωφέλη σε ένα τομέα πολιτικής μπορούμε να έχουμε ωφέλη και σε άλλους τομείς πολιτικής. Φυσικά υπάρχουν και άλλα τομείς που θα πρέπει να διερευνήσουμε και αν δούμε ε, και την ε, βασική νομοθεσία και με τη ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ ε, Enterprise όταν εξετάσουμε τα πρότυπα για τα αυτοκίνητα που καίνε diesel και να αξιολογήσουμε και αυτή τη διαδικασία σε συνδυασμό με αυτή εδώ. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να προκύψουν και από εκεί ωφέλη και νομίζω ότι είναι σημαντικό όταν θέτουμε φιλόδοξους στόχους όπως μας δείξατε πολύ καλά να μην ε, αυξάνουμε το κόστος με όρους πολιτικής και να μπορούμε το ίδιο να το επαναλάβουμε και για άλλους τομείς. Ε, και για τα επόμενα πρότυπα, για τα αυτοκίνητα diesel, θα συνεργαστούμε που σας είπα πολύ στενά και με τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να δώσω το λόγο στην κρυφαρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρους της κυρίας Κάθριν Παιδί που είναι σκιώδη εισηγήτρια από την ομάδα των φιλελευθέρων και δεδομένη της παρουσίαση της μελέτη αντικτύπου για τις προτάσεις της Κομισιόν, θέλω να θέσω την εξή ερώτηση. Ο Γεωργικός τομέας έχει συνεισφέρει για πολύ καιρό ε, στι εκπομπέ στην ατμόσφαιρα. Κύριος, ε, κύριε Μάρκου Σάμεν όταν ε, κάνατε αυτή τη μελέτη δικτύπου, συναντήσετε κάποια στοιχεία σε σχέση ε, με το πόσο θα συνεισφέρει ο γεωργικός τομέας για να πετύχουμε το κόστος για το μεθάνιο για το 2030 και μπορείτε να μας πείτε πόσο ακριβώ θα επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Η κυρία Κονέτσα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω τους συντάκτες της ε, μελέτης που δείχνουν ποια πορεία πρέπει να ακολουθήσουμε. Και νομίζω ότι τη μελέτη αυτή οφείλουμε να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη. Γιατί αυτό το λέω διότι ορισμένες από τις οδηγίες μας επικαλύπτονται αλλά δεν αναπτύσσονται οι απαραίτητες συνέργειες και συχνά η μία καταμάχεται την άλλη στα αποτελέσματα. Νομίζω λοιπόν ότι όντως χρειάζεται να γνωρίζουμε τους αντικτύπους του κάθε νομοθετήματος για να συνεχίσουμε την εργασία μας. Εγώ βλέπω με ικανοποίηση ότι οι, στόχοι, οι κλιματικοί στόχοι του Συμβουλίου είναι θετικοί σε ό,τι αφορά τον καθαρό αέρα και αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση για μείωση των εκπομπών. Εκτιμώ την προσπάθεια να περιληφθούν και πολύ συγκεκριμένα πράγματα όπως ανώτατες τιμές για στερεά σωματίδια. Από την άλλη μεριά, μιλώντας για το μεθάνιο, έχω να πω ότι ίσως δεν είναι απαραίτητο να είναι η πρώτη προτεραιότητα για μας. Ίσως έχει κάποια σημασία για τη γεωργία. Αλλά στα πλαίσια των υπόλοιπων μέτρων μας, το μεθάνιο, ας μη θεωρηθεί τόσο σημαντικό. Που να αξίζει να εγκύψουμε σε ειδικέ λύσεις γι' αυτό. σε μια προσπάθεια να μειώσουμε και άλλες ουσίες. Επίσης οι εκπομπές αμμονίας πρέπει να μειωθούν όπως άλλωστε δείχνουν τα σχεδιαγράμματα, οι γραφικές παραστάσεις που μας έδειξαν. Και εκεί κάτι πρέπει να κάνουμε. Ας μην λησμονούμε πάντως τους τελικούς στόχους μας. Να αποφύγουμε τις επικαλύψεις δηλαδή και να προβούμε στις περιορισμούς που είναι απαραίτητοι. Eichhout. Ευχαριστώ πρώτα τον Μάρκους Άμαν για την δουλειά και την ξεκαθαρή παρουσίαση. Γνωρίζοντας άλλωστε ότι ο προϋπολογισμός της μελέτης αλλά και ο διαθέσιμος χρόνος δεν ήταν άφθονα. Ξέρω ότι δουλέψατε και στις διακοπές σας και γι' αυτό νομίζω ότι οφείλουμε να εκτιμήσουμε ιδιαίτερα τη δουλειά που κάνατε. Και που δείχνει άλλωστε ότι πρέπει να περιληφθούν και οι διασυνδέσεις μεταξύ του τι κάνουμε από τη μια μεριά για το κλίμα και την ενέργεια και από την άλλη μεριά για την ποιότητα του αέρα. Η μελέτη δείχνει αυτούς τους συσχετισμούς αλλά και τα παρελκόμενα ωφέλη από τις πολιτικές αυτές. Πρώτη ερώτηση θα κάνετε και μια παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης σας στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. Κάτι τέτοιο αξίζει τον κόπο γιατί γνωρίζουμε ότι εντός των κόλπων του Συμβουλίου τους ενδιαφέρουν ιδίω να, τα αποτελέσματα του κόστους του κάθε νομοθετήματος και όχι τα αποτελέσματα στην υγεία κτλ. Συνήθως οι συζητήσεις στο Συμβούλιο περιορίζονται στην μελέτη του κόστους. Θα έπρεπε να τους δείξουμε και ποια είναι τα ωφέλη για την υγεία και ιδίω σε συνδυασμό με τις πολιτικές ενέργειας και κλίματος, στις οποίες, τις οποίες έχουν προσυπογράψει οι χώρες μέλη, βέβαια με κάποιες αποκλήσεις και με κάποιες άλλες πονηριές, αλλά τουλάχιστον να γίνει συζήτηση και στο Συμβουλίο, έτσι ώστε να μετακινηθεί κάπως η προσοχή τους και η στόχευσή τους από το, στόχος, από το κόστος μονάχα. Άλλωστε η μελέτη σας δείχνει, και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, ότι εάν εξετάσουμε την, αν προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τις άκρες ανάμεσα σε αυτό που είναι τεχνικά δυνατό και στα άλλα αποτελέσματα η Κομισιόν είπε ότι για το 67%, 67% και ήδη γι' αυτό μπορεί να επικριθεί διότι είναι πάρα πολύ συντηρητική η εκτίμησή της. Αν δείτε την ε, baseline, την βάση η καλύτερη προσέγγιση ήταν μεταξύ 76% και 92%. Ήδη λοιπόν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι υπερβολικά συντηρητική. Αν περιληφθούν τώρα και τα άλλα συν ωφέλη, πρέπει πάλι να εξεταστεί με τον τρόπο αυτό η πρόταση της Επιτροπής και είναι σαφές για τα άλλα θεσμικά όργανα και για το Συμβούλιο, γιατί πάντα μιλούν για πολιτικές βασισμένες σε γεγονότα, σε επιστημονικά δεδομένα. Δείχνει όμως η μελέτη καθαρά. Επιτέλους τι συζητούμε τότε αρχίζει και γίνεται αστείο αυτό. Βέβαια, την ερώτηση αυτή τη διαβιβάζω ιδίω προ τα άλλα θεσμικά όργανα. Δεν είναι ερώτηση προ εσά, είναι και πολιτική η δήλωσή μου. Εσεί είστε επιστήμον και βεβαίω απέχετε από οποιασδήποτε ε, πολιτικέ δηλώσει. Και σωστά κάνετε. Τελευταία ερώτηση τώρα, αν, εκτός από το αν θα πάτε στο Συμβούλιο να κάνετε την παρουσίαση, όταν συζητούμε και άλλες ε, τροπολογίες για την πρόταση της Επιτροπής, θα χρειαστούμε και δεδομένα αναχώρα. Εγώ γνωρίζω ότι στο μοντέλο που καταστρώνεται θα πρέπει να υπάρχει και το κόστος της μείωσης των εκπομπών αναχώρα. Μπορείτε να μας δώσετε σχετικά δεδομένα, σχετικά στοιχεία. Το άλλο είναι βέβαια τα ωφελήματα για την υγεία αναχώρα. Πιθανώς θα χρειαστεί και άλλη ανάλυση και όχι μόνο από δική σας πλευρά αλλά και κάποια συνεργασία ίσως με τον Μάικ Χόλαντ. Είναι δυνατόν λοιπόν να έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα για τα ωφέλη στην υγεία αναχώρα. Τελευταία ερώτηση. Έχετε και δεδομένα για το 2020, γιατί αυτό θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Και επειδή μιλείτε ήδη για 2025 και 2030, θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται και το 2020. Ευχαριστώ, ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για αυτή την παρουσίαση και εμείς ε, θα μελετήσουμε εις βάθος τη μελέτη αντικτύπου. Εδώ έχουμε μία πρόταση να κάνουμε. Η πρόταση οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα ορίζει νέε δεσμεύσει μείωση ε, για τι ε, κάποιες ε, εκπομπές διοξιδίου του θείου, οξιδίου του αζότου και αμμονία και μεθανίου. Όμως ε, δεν έχουμε ε, το... τα νητρικά άλατα είναι πάρα πολύ επιζήμια και έχουμε 0,001 σωματίδια ένα εκατομμύριο ενώ ε, αν ε, είμαστε κοντά σε δηληστήρια έχουμε 3,3 μέρη ανά εκατομμύριο. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε πολλές φορές περισσότερο πολύ περισσότερα τέτοια σωματίδια. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ αρνητικές οι επιπτώσεις, αλλά δεν γνωρίζουμε τις επιπτώσεις της χρόνιας έκθεσης του πληθυσμού που ζει κοντά στα δηληστήρια. Έτσι λοιπόν εμείς προτείνουμε να διευρύνουμε τον κατάλογο για το υδρογονωμένο ε, φόσφορο που είναι και μία αιτία που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Σας ευχαριστώ. Καρθάινς Φλόρενς. Κοιτάξτε, πολλές ερωτήσεις έχουν ήδη υποβληθεί Θα ήθελα να μου πείτε αν έχει υπάρξει αντίδραση της Κομισιόν. Εάν υπάρχει ε, ενδεχόμενο τροποποίησης της στρατηγικής. Κοιτάξτε, για το κόστος πάντα εμένα με κάνει φιλίποπτο όταν ε, λέμε ότι όλα αυτά έχουν ε, μηδενικό κόστος. Φυσικά από πλευράς μιας σφαιρικής αντιμετώπισης μπορεί να είναι εποφελή, αλλά αν είναι κανείς επιχειρηματίας ή γεωργός ε, τα βλέπει κάπως διαφορετικά. Μπορείτε να μας πείτε εάν ε, έχετε κάποια στοιχεία για τη γεωργία για να μην με εκτελέσουν αύριο που θα πάω στην εκλογική μου περιφέρεια να μιλήσω στους γεωργούς. Δεν ξέρω αν είναι δυνατόν να πω συγκεκριμένα, αλλά μια ιδέα. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Γκρότε. Αυτό που είπε ο Άικχαουτ νομίζω ότι είναι σωστό. Αυτά πρέπει να τα πείτε και στο Συμβούλιο. Αν δει κανεί πώς έχει η αντιμετώπιση του κλίματος με βάση τα πορίσματα του Οκτωβρίου, θα ήταν πολύ χρήσιμο να είχαν αυτά τα στοιχεία όταν τα συζήτησαν. Πολλά ήδη αναφέρθηκαν. Το θέμα είναι Εάν συνδέσει κανείς τα ωφέλη για την υγεία με την προστασία του περιβάλλοντος, δεν είναι εύκολο να εξηγήσει κανείς. Γιατί αν τους πούμε ότι για την προστασία του κλίματος πρέπει να χαθούν θέσεις εργασίας, δεν θα κερδίσει εκλογές ποτέ. Αλλά, εν περιπτώσει, είναι πολύ ουσιώδες αυτό που λέτε, ότι θα αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής κατά 4,4 μήνες, αλλά αυτά τα στατιστικά στοιχεία είναι δυσνόητα για τον απλό πολίτη. Η ερώτησή μου, ε, σε τι βαθμό υπολογίσατε και πιο αισιόδοξου στόχους. Βασιστήκατε μόνο σε αυτά που έχουν ήδη κατατεθεί και είναι επιτάπητος. Θα με ενδιέφερε να μου πείτε εάν υπολογίσατε πόσο υψηλότερα θα ήταν τα ωφέλεια αν είχαμε πιο αισιόδοξου στόχους. Ε, είναι πραγματικά εντυπωσιακή όμως ε, γενικότερα η μελέτη σας. ευχαριστώ πολύ και να δούμε εάν θα μπορούσαμε να την αποστείλουμε και στα άλλα δύο θεσμικά όργανα. Θαυμάσια εργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πριν να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Αμάν για να απαντήσει, εγώ θα ζητούσα από την Κομισιόν να πάρει το λόγο αν θέλει να σχολιάσει τη μελέτη αυτή. Γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντική και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, όντω είναι σημαντική. Καταρχήν, εκ μέρους Κομισιόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Επιτροπή σα, επειδή έχουμε πρόσθετα αριθμητικά στοιχεία, γιατί είναι μια πολιτική που θα μπορούσε να είναι αρκετά πολύπλοκη, αλλά αυτό τονίστηκε και στην, ε, να έχει μάλλον στοιχειοθετηθεί. Από εκτατική, εκτεταμένη ανάλυση στην πρόταση της Κομισιόν, νομίζω ότι εδώ είμαστε μαζί σας για να μάθουμε για να ακούσουμε και φυσικά αυτό πράττουμε. Πραγματικά είναι εύκολο να χαθεί κανεί ε, σε όλα αυτά τα αριθμητικά στοιχεία, όπω είπε και ο συγητή. Και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια επιπλέον για να καταλάβουμε ε, όλα αυτά τα στοιχεία και αυτό θα μας βοηθήσει και στις διαπραγματεύσεις. Όμως τώρα να υπενθυμίσω τι έκανε η Κομισιόν τότε, η πρόταση της Κομισιόν. Ουσιαστικά παρουσίαζε μια πρόταση ΝΕΚ για τα εθνικά όρια εκπομπών, αλλά ο έσχατος στόχος ή το έσχατο αποτέλεσμα θα ήταν να μειώσουμε τους πρώιμους θανάτους από την ατμοσφαιρική ρήπανση. Σήμερα έχουμε περίπου 400.000 τέτοιους θανάτους ετησίως. Να το μειώσουμε λοιπόν αυτό το επίπεδο θανάτων και να φτάσουμε στις 200.000. Από την παρουσίαση αυτή, τι κρατάμε. Ότι μπορεί κανείς να κάνει περισσότερα με το ίδιο ποσό, χρημάτων ή το ίδιο με λιγότερα χρήματα. Υπάρχουν πάρα πολλέ ενδιαφέρουσε πληροφορίε λοιπόν επιτάπητο. Είμαι σίγουρο ότι θα τροφοδοτήσουν τι διαπραγματεύσει και φυσικά θα έχουμε υψηλότερη ποιότητα διαπραγματεύσεων ή τουλάχιστον έτσι ελπίζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τι πληροφορίε αυτέ ε, που τι συνεισφέρετε στη συζήτηση. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να δώσω το λόγο στον καθηγητή Αμάν για να απαντήσει τις ερωτήσεις που έκανε οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα δώσω κάποιε σύντομε απαντήσει. Υπήρχε μια ερώτηση για τι εκπομπέ ε, του μεθανίου και το κόστο ε, των προτινόμενων μέτρων για το μεθάνιο, ιδίω στον τομέα τη γεωργία. Είναι σαφέ ότι το μεθάνιο είναι σίγουρα ένα αέριο του θερμοκηπίου και φυσικά αποτελεί τμήμα του πακέτου κλίματος και ενέργειας και η συζήτηση έχει να κάνει με το αν είναι στο σύστημα εμπορίας θα υπάρχει φυσικά κάποια τιμή ε, για τον άνθρακα. Ανάλογα με το πώς θα καθοριστεί η τιμή αυτή. Το νέο στοιχείο εδώ είναι ότι η πρόταση αναγνωρίζει το μεθοανείο και ως ατμοσφαιρικό ρήπο Πρόκειται για μια σημαντική πρόδρυμη ουσία ε, του όζοντος ε, που δεν έχει αναγνωριστεί επιστημονικά προηγουμένως, αλλά συνεισφέρει ε, σε αυτό, στο όζον που βλάπτει την ανθρώπινη υγεία, δηλαδή βλάπτει και την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Η πρόταση της Κομισιόν είναι να λάβει τα μέτρα που θα μπορούσαν να επιτευχθούν με μηδενικό κόστος. Έχουμε φυσικά τις αρχικές επενδύσεις ε, που καλύπτονται με κατόπιν εξοικονομήσεις. Ε, έχουμε δηλαδή μια αρχική επένδυση για ε, το βιοαέριο, αλλά κατόπιν μπορούμε να έχουμε εξοικονόμηση. Έτσι λοιπόν η πρόταση της Κομισιόν προτείνει για στόχους ποιότητας του αέρα να πάρουμε αυτά τα μέτρα για το μεθάνιο που δεν έχουν κόστος. Έτσι λοιπόν η απάντηση στην ερώτηση είναι ότι το κόστος για το μεθάνιο και για την τομέα της γεωργίας είναι μηδενικό στην πρόταση της Κομισιόν. Τώρα η, πρόταση, η κλιματική πρόταση είναι πιο φιλόδοξη. Υπήρχε και άλλη μια ερώτηση σχετικά με το αν έχουμε στοιχεία ε, για τα ωφέλη της υγείας και για το κόστος. Δεν υπάρχουν στο έγγραφο, αλλά εύκολα θα μπορούσαμε να σας τα διαθέσουμε και στο διαδίκτυο. Όλες αυτές τις πληροφορίες υπάρχουν στο διαδίκτυο, διαθέσιμες. Μπορείτε στην ιστοσελίδα να βρείτε όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Και τα δεδομένα υπάρχουν και για το 2020 επί της αρχής, αν και δεν είχαμε χρόνο να τα κυρώσουμε και να συζητήσουμε με τους εθνικούς εμπειρογνώμονες τα εθνικά δεδομένα. Υπάρχει ε, λοιπόν ε, ε, ένα πρόβλημα με αυτά τα δεδομένα γιατί δεν είχαμε χρόνο να τα εξετάσουμε λεπτομερώς. Ο μακροοικονομικός αντίκτυπος. Ναι, έχει αναλυθεί εκτενώς ποιος θα είναι ο αντίκτυπος της πρότασης ε, και ε, η ροή χρημάτων πίσω στην οικονομία. Υπήρχε και μια συγκεκριμένη πτυχή για την κατανομή του άχθους σε διάφορους τομείς, τον επιμερισμό του άχθους. την ε, βέλτιστη οικονομική προοπτική, την πρόταση της Κομισιόν, ε, είχαμε κλείσιμο του χάσματος 60, ε, συγγνώμη, 75% και εξετάσαμε τι συμβαίνει και με το άφθος στο γεωργικό τομέα. Και αυτό ήταν ένα από τα επιχειρήματα της Κομισιόν για να περάσουμε από το 75% στο 67%. Όμως μπορούμε να πούμε ότι αυτό το άχθος ε, στο γεωργικό τομέα θα προκύψει μόνο αν δούμε το πρόσθετο κόστος. Αν ε, δούμε τι πληρώνουν τώρα οι βιομηχανίες με τη σημερινή νομοθεσία, ε, το κόστος για τη γεωργία είναι πολύ χαμηλό. Κυρίως το κόστος το πληρώνει η βιομηχανία, ο τομέας των μεταφορών, τομέας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι λοιπόν υπάρχουν πολύ ε, μεγάλες αποκλήσεις ε, σε σχέση με το κόστος που καταβάλει ο κάθε τομέας. Το κύριο άχθος το έχει η βιομηχανία, ο τομέας των μεταφορών όπως σας είπα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, πολύ μικρό το κόστος για τη γεωργία. Στη νέα πρόταση ε, καλύπτει κάπως και η γεωργία και εξισορροπείται κατά κάποιο τρόπο το κόστος αν ε, δείτε τι συμβαίνει στο περιθώριο, ε, θα δείτε ότι υπάρχει αύξηση του κόστους για τη Γεωργία, αν δείτε όμως το συνολικό παραμένει πολύ χαμηλό. Και υπήρχε και μία ερώτηση για το αν έχουμε αναλύσει πιο φιλόδοξους στόχους, ναι. Έχουμε αναλύσει την πλήρη γκάμα από το 0% στο 100%, 100% ε, με συγχωρείτε, και με το 5% ενδιάμεσα. Βέβαια, ε, εξαφανίστηκαν ε, πολύ γρήγορα από τη συζήτηση πιο φιλοδεξιτόχοι και επικεντρωθήκαμε σε αυτά που είδατε στην πρόταση. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Μπορούμε τώρα να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, δίνοντας το λόγο στον εισηγητή. Um, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή ορισμένα που θέλω να πω. Ως εισηγήτρια βέβαια ασχολήθηκα κάπως περισσότερο με το θέμα αυτό. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό που συζητάμε είναι μία οικονομική μελέτη με βάση ορισμένες προϋποθέσεις και δέχομαι απόλυτα ότι θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε μια κάπως διαφορετική προσέγγιση από την πρόταση της Κομισιόν, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι οι μεταβλητές βάσει των οποίων εκπονήθηκε δεν είναι απόλυτα σίγουρες. Έχουμε για παράδειγμα μία εκτίμηση για την οικονομική ανάπτυξη από τώρα μέχρι το 2030 και άλλες μεταβλητές, το κόστος του άνθρακα και κάτι πολύ σημαντικό που δεν νομίζω ότι προέκυψε από τη συζήτηση. Τα διάφορα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο για τα εθνικά όρια εκπομπών, δηλαδή οι διάφοροι ρήποι, μιλήσαμε για την αμμονία και το μεθάνιο και το πώς επιδρούν στη γεωργία. Δεν ε, έχουν ε, ισότιμο βάρος από πλευρά συμμετοχής τους στα αέρια θερμοκηπίου. Το καθένα ε, παίζει διαφορετικό ρόλο. Βεβαίως λοιπόν ε, όταν εξετάζουμε το συνολικό πλαίσιο για τις εθνικές εκπομπές θέλουμε να καθορίσουμε ένα συνολικό φιλόδοξο όριο αλλά ορισμένες πολιτικές δεν αμφισβητούνται ορισμένες εθνικές πολιτικές δεν μπορούμε να τις αγνοήσουμε ορισμένες πολιτικές ιδιαίτερα για τις πρώτες ύλες θα επιδράσουν επί των ρηπαντών και θα πρέπει να δούμε εάν το μοντέλο που προτείνουμε έχει τελικά έννοια. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Διότι ναι μεν εμείς εδώ δεν αμφισβητούμε ε, το μοντέλο αυτό. Ξέρω ότι πολλοί θα απευθυνθούν και σε μένα και στους κοιόδης για να το αμφισβητήσουν. Πρέπει λοιπόν να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι θέλουμε να βασίσουμε τις συζητήσεις μας Εάν θέλουμε να συζητήσουμε, να, συγγνώμη, να βασίσουμε τις συζητήσεις μας πλήρως σε αυτό, βεβαίως αυτή η μελέτη κόστους ωφέλους, αυτό το περιθωριακό κόστος αλλάζει ανάλογα με το τι δράσεις θα υιοθετήσουμε. Αλλά όσο προχωράμε, μοιάζει να είναι προφανές ότι αυτό πρέπει να κάνουμε, αυτό πρέπει να έχουμε πιο φιλόδοξους στόχους για να επιτύχουμε περισσότερα ωφέλη, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε πολύ πιο προσεκτικά. Τι εννοώ λοιπόν. Εγώ θα συζητήσω και με την Επιτροπή αναλυτικά για να δω πώς θα αντιδράσει. Γιατί η αρχική αντίδραση ήταν κάπως γενικόλογη, όπως την ακούσαμε από τους εκπροσώπους της Κομισιόν. Πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες και να δούμε πού θα μας πάνε οι λεπτομέρειες. Και συμφωνώ απόλυτα αυτό που είπατε ότι και το κόστος και το όφελος ε, μπορούν να αφορούν διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, άρα δεν φαίνονται πλήρως από μια πρώτη γενική ματιά και το 2030 απέχει πολύ, μπορεί να αλλάξουν στόχοι της πολιτικής. Πρέπει λοιπόν στο πλαίσιο αυτό των στόχων NEC, δηλαδή ε, εθνικών ε, ανώτατων ορίων για τους ρηπαντές, να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί. Τι θα ήθελα λοιπόν να πω σε όλους μας και κυρίως στους Κιώδης. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη για αυτό το θέμα. Πρέπει να κάνουμε πολλές αναλύσεις, να συνεργαστούμε πολύ για να διασφαλίσουμε ότι θα καταλήξουμε σε κάτι συνενετικό. Η έκθεση αυτή είναι πολύ χρήσιμη που ακούσαμε και όπως είπα θα συζητήσω και με την αντίστοιχη υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη μελέτη κατά τις συζητήσεις μας για να δούμε σε ποιο επίπεδο μπορούμε να θέσουμε τις φιλοδοξίες μας. Ευχαριστώ πολύ τη συνάδελφο Γκίρλινγκ που είναι η συγγήτριά μας για τα Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό και να παράσουμε στο επόμενο. Όπως θα θυμάστε, όταν εγκρίναμε την ημερήσια διάταξη, για τη συνεδρίασή μας. Αντιστρέψαμε τα 18-19, οπότε τώρα θα μιλήσουμε για την απαγόρευση αλληλείας με παρασυρώμενα δίχτυα. Όπως ξέρετε, ο κανονισμός που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει την απαγόρευση αυτών των δικτύων λόγω της αρνητικής επίπτωσής τους επί του περιβάλλοντος, λόγω των παραπλεύρων αλλιεμάτων από αυτά τα δίκτυα και, και δίνω αμέσως το λόγο στον κύριο Αφρόντε που είναι ο εισηγητής μας. Παρακαλώ. Παρακαλώ όμως επίσης συνάδελφοι όσοι αποχωρούν να αποχωρήσουν χωρίς φασαρία διότι οι εργασίες της Επιτροπής μας δεν έχουν διακοπεί, συνεχίζονται. Ο κύριος Αφρόντε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λοιπόν, τα παρασυρώμενα δίχτυα είναι αλληλευτικά εργαλεία με τον οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολύ. Είναι τα δίχτυα που μπορεί να ε, φτάνουν μέχρι και εκατοντάδες μέτρα. Αυτή τη στιγμή απαγορεύονται στα ευρωπαϊκά δίκτυα. Ε, δίχτυα πάνω από 2,5 χιλιόμετρα. Έτσι λοιπόν αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποια σκάφη να έχουν πάρα πολύ μακριά δίχτυα. Έτσι λοιπόν ε, καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα τεράστιο αντίκτυπο αυτών των δίχτυων στο περιβάλλον. Από τη δεκαετία του 90 αυτά τα δίχτυα να έχουν μεγάλο μάτι και η διεύρυνση των ματιών οδήγησε σε έναν αντίκτυπο σε ορισμένα προστατευόμενα είδη που είναι και υψηλά μεταναστευτικά είδη που είναι και πάρα πολύ σημαντικά για την προστασία ε, των ειδών. Μιλάμε για τα δελφίνια, για τους καρχαρίες, ε, για τον ξηφία. Η πρόταση της Κομισιόν γεννάται και σε ένα πολύ ιδιαίτερο πλαίσιο γιατί η ίδια η Κομισιόν ε, μας ε, λέει στην περίληψη της πρότασής της ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη νομοθετική κατάσταση. Η ίδια η Κομισιόν αναφέρει ότι ε, μπορεί κάποιος να παρακάμψει εύκολα την ισχύουσα νομοθεσία και υπογραμμίζει ότι επέτρεψε αυτή η νομοθεσία να ε, ε, μπορούν να χρησιμοποιούν οι αλείς παράνομα αυτά τα δίκτυα που έχουν απαγορευτεί και λέει ότι παρόλα αυτά, παρά την ισχυρή νομοθεσία, στα ίδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζουμε να βλέπουμε παράνομη χρήση αυτών των παρασυρώμενων δικτυών. Υπήρχαν και δύο αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εναντί της Γαλλίας και της Ιταλίας. Και σε αυτό το ιδιαίτερα πολύπλοκο πλαίσιο και μπροστά σε ένα αλληλευτικό εργαλείο που έχει ένα πολύ μεγάλο αντίκτυπο και στο περιβάλλον και στα προστατευόμενα είδη, η Κομισιόν έκανε μία πρόταση που πολλοί θεώρησαν ότι είναι προκλητική. Μία πρόταση η οποία ουσιαστικά έχει μια πολύ σκληρή γραμμή. Δηλαδή λέει να απαγορεύσουμε σε όλα τη δε της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη χρήση των παρασυρώμενων δικτυών. Αναφέρει τέσσερα άρθρα μόνο και το άρθρο 3 είναι πολύ σημαντικό και λέει ότι απαγορεύεται σε όλα τα ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να χρησιμοποιούνται αυτά τα δίκτυα και να υπάρχει οποιοδήποτε είδους ε, τέτοιο παρασυρώμενο δικτυού επάνω στα σκάφη. Για να φτάσουμε στην πρόταση αυτή, για να φτάσει στην πρόταση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προφανώς προετοίμασε μια μελέτη αντικτύπου στην οποία τα σημεία και οι επιλογές που είχε κατά νου ήταν τέσσερα. Καταρχήν να διατηρήσει τη σημερινή κατάσταση τόσο κράτους ΒΟ μέχρι την τελευταία που ήταν η ολική απαγόρευση της χρήσης αυτών των δικτυών. Στη μέση υπήρχαν και κάποιες εναλλακτικές, μία από αυτές ε, δηλαδή η τιμία θα την αναφέρω, γιατί θα επαναφέρουμε, σε αυτό το θέμα. Δηλαδή να έχουμε επιλεκτική απαγόρευση, να βρούμε ποια είναι αυτά τα δίκτυα που είναι τα πιο επικίνδυνα και έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο για το περιβάλλον και να χτυπήσουμε μόνο εκείνα τα είδη δικτυών. Βέβαια το πρόβλημα είναι ότι στην ίδια τη μελέτη αντικτύπου για αυτή την τρίτη επιλογή που πιθανότητα μάλλον θα άρεσε περισσότερο ίσως και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι μόνο στις επιτροπές που αναλύουν αυτή και πρόκειται για την Επιτροπή Ελίας πέρα από τη δική μας, στην ίδια τη μελέτη αντικτή που λέει η Κομισιόν. Εντάξει, η επιλογή τρία είναι η επιλεκτική απαγόρευση, όμως ε, προς στιγμή δεν έχουμε πληροφορίες που να μας επιτρέπουν με ακρίβεια να δούμε ποιε είναι οι πιο επιζήμιες δραστηριότητες, έτσι λοιπόν θα ήταν καλύτερο να συνεχίσουμε τις έρευνες στον τομέα αυτό. Η επιλογή 3, δηλαδή επιλεκτική απαγόρευση, είναι μια καλή επιλογή, όμως δυστυχώς δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να μπορέσουμε να την προωθήσουμε και να τις προσδώσουμε συνέχεια. Βάση λοιπόν ενός ε, δύσκολου ρυθμιστικού πλησίου περμηνευτική σκοπιά και το οποίο δυστυχώς ε, παραβιάζεται πάρα πολλές φορές και κάτι που θα μπορούσε να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά τελικά δεν το έκανε γιατί δεν έχει στοιχεία, φτάνει η Κομισιόν στο να προτείνει την πλήρη απαγόρευση τη αλληλεία με παρασυρωμένα δίχτυα. Αυτή η αιωλική απαγόρευση ε, και για τα ενδιαφέρα μέρη, αλλά και στις πρώτες συζητήσεις που είχαμε στην Επιτροπή Αλία, συνάντησε πάρα πολύ ισχυρέ αντιδράσεις και διάχυτες και σε επίπεδο των ενδιαφερομένων μερών, αλλά και σε επίπεδο πολιτικών ομάδων που συζητούν στην Επιτροπή Αλίας. Οι κύριες αντιρρήσεις είναι τρεις. Η πρώτη είναι ότι η διάταξη δεν λαμβάνει υπόψη έναν ε, βασικό πυλώνα της ε, κοινή ελευτικής πολιτικής, δηλαδή την περιφερειοποίηση, δηλαδή το γεγονό ότι τα μεμονωμένα κράτη πρέπει να εκτιμήσουν την τοπική κατάσταση και να λάβουν μέτρα. Δεύτερη περίοδος ότι θα χτυπούσε η νομοθεσία κάποιες μικρές κοινότητες αλληλευτικές που πράγματι χρησιμοποιούν κάποια τέτοια είδη δικτυών παρασυρώμενα που όμως δεν έχουν και πολύ μεγάλο αντίκτυπο στο περιβάλλον, έχουν μάλλον μικρό αντίκτυπο και κάτι άλλο σημείο που είπαμε, κάποιο άλλο σημείο που είπαμε ήδη, ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε η αντίκτυπο θα είχε μια επιλεκτική απαγόρευση. Επίση έχουμε το πρόβλημα και του ορισμού. Εγώ στην γνωμοδότησή μου έχω προτείνει έναν ορισμό, δηλαδή να θέσουμε σε εφαρμογή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ορισμό, καθώς είναι κάπως πιο διευρυμένος, αλλά αυτό είναι ένα τεχνικό στοιχείο. Και ερχόμαστε τώρα και στην πρόταση γνωμοδότησης για να μπορούμε να διατυπώσουμε μία πρόταση γνωμοδότηση στην περίπτωση αυτή, δεδομένου ότι η πρόταση τη Κομισιόν είναι πράγματι πολύ συγκεκριμένη, πολύ σύντομη, ξεκάθαρη, πλήρης απαγόρευση. Αλλά θέλοντας να απαντήσουμε στις αντιρρήσεις των ενδιαφερομένων μερών και των συναδέλφων της Επιτροπής Ελίας, και όπως σας είπα, αντιρρήσεις ε, προήλθαν ε, σχεδόν ε, από όλες τις πολιτικές ομάδες. Εγώ έλαβα υπόψη αυτές τις αντιρρήσεις και προσπάθησα να βρω μια εναλλακτική. Η πρότασή μου λοιπόν, που θέτω εδώ σήμερα προς δική σας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, είναι η εξή. Να αφήσουμε τα κράτη-μέλη να λάβουν την απόφαση. Έτσι λοιπόν, σε εκείνο το σημείο θα βρουν μία διπλή οδό. Καταρχήν, κάθε κρατούν μέλος μπορεί αυτόνομα να αποφασίσει, να προχωρήσει και να προβεί σε πλήρη απαγόρευση των παρασυρώμενων δικτυών ή αν αποφασίσουν να μην προβούν στην ολική απαγόρευση, θα μπορούσαν να ακολουθήσουν η άλλη οδό που να τους επιτρέπει κατά παρέκκληση αυτής της απαγόρευση να χρησιμοποιούνται, να επιτρέψουν να χρησιμοποιούνται τα δίχτυα περίπου για ένα εναμιση χρόνο ακόμη μέχρι τα μέσα του 2017 και στην περίοδο αυτή θα πρέπει να απαντήσουν τις απαιτήσει που έχουν προκύψει, δηλαδή στο ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία. Δηλαδή μπορούν κατά παρέκκληση να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν αυτά τα δίκτυα, αλλά θα πρέπει εντωμεταξύ να συλλέξουν μία σειρά στοιχείων. Θα πρέπει να κάνουν ένα κατάλογο των διάφορων ειδών δικτυών που χρησιμοποιούνται, να αξιολογήσουν για κάθε είδους δικτυού ε, ποια είναι, ποιος είναι ο ακριβής αντίκτυπος που έχει το κάθε μεμονωμένο λευτικό εργαλείο, ιδιαίτερα για τα είδη που αναφέρονται για τα προστατευόμενα είδη και για τα ιδίω μεταναστευτικά είδη, μελέτη σε βάθος για το πιο αντίκτυπο θα είχε η απαγόρευση αυτών των δικτυών στις κοινότητες, δηλαδή από κοινωνική και οικονομική σκοπιά. Και επίση, στο τέλος αυτής της καταπαρέκκληση περιόδου, θα πρέπει να παρουσιαστούν όλα αυτά τα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αφού θα αξιολογήσει όλα αυτά τα στοιχεία. Και χρησιμοποιώντας όσο δυνατό πληρέστερα κριτήρια, εκ νέου θα έχει κομισιόν στα χέρια της τη δυνατότητα να απαγορεύσει επιλεκτικά αυτά τα παρασυρώμενα δίκτυα. Δηλαδή θα αξιολογήσει ποια είναι ακριβώς τα εργαλεία που έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο στο περιβάλλον και πρέπει να απαγορευτούν, ενώ για κάποια άλλα δίκτυα, για λογικούς και οικονομικούς λόγους θα μπορούσε να επιτραπεί να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται. Σα καλώ όλου να αξιολογήσετε αυτή τη γνωμοδότηση έχοντα κατά νου ότι Καθώ πρόκειται για μια εναλλακτική σε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση αναγκαστικά μα απομακρύνει αρκετά από την αρχική πρόταση τη Κομισιόν. Όμω, καθώ βρισκόμαστε ενώπιον μια επιλογή μεταξύ του να υιοθετήσουμε την πλήρη απαγόρευση των περασυνόμενων δικτυών ω έχει και από ό,τι φαίνεται σε όλα τα μέρη και σε όλες ε, τις ομάδες ε, δεν φάνηκε κάτι αποδεκτό, πρέπει να βρούμε μια εναλλακτική που να μας επιτρέπει όμως να ακολουθήσουμε την κύρια οδό, δηλαδή να εξυπηρετήσουμε τον κύριο μας στόχο να απαγορεύσουμε τελικά τα δίθια που έχουν ένα πολύ μεγάλο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Αυτό είναι ο κύριος στόχος, το υπενθυμίζω. Και με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και αν θα έχουμε μεγαλύτερες προθεσμίες, το λέω αυτό δυστυχώς, γιατί πάντα δεν είναι πλέον έκτημα αυτό, αφήσουμε και μία πρωτοβουλία στα κράτη-μέλη, αλλά θα αφήσουμε και τη δυνατότητα στις μικρές αλληλευτικές κοινότητες να συνεχίσουν το έργο τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Σίγητη για την παρουσίαση αυτή. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στους κοιόδης εισηγητές. Ξεκινήσουμε με το ΕΛΚ από την κυρία Ράνς Γκαρσία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταργηθούν ε, από τη μια μέρα στην άλλη όλα τα παρασυρώμενα δίκτυα μας εξέπληξε. Διότι Ορισμένα από αυτά τα δίκτυα ε, δεν προκαλούν καμία βλάβη στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, η αλία της Σαρδέλα στην Γαλλικία όπου χρησιμοποιείται ένα συγκεκριμένο είδος δικτυών είναι μικρής κλίμακας και ασχολείται μόνο με τη σαρδέλα αναπτύσσεται, λοιπόν γίνεται αυτή η δραστηριότητα χωρίς να προκαλεί ζημία σε απειλούμενα είδη και χωρίς να αλλιεύει είδη που δεν επιτρέπονται. Άρα δεν είναι δυνατόν να απαγορεύσουμε αυτά τα δίκτυα. Και καταλαβαίνετε ότι θα προκαλούσε σημαντική κοινωνικο-οικονομική ε, ζημιά σε 400 περίπου σκάφη. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την πρόταση λοιπόν. Κοιτάξτε, είναι σαν να σκοτώνουμε μύγες με κανόνια. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο πονάει δόντι κόβει κεφάλι. Χωρίς να αντιμετωπίζουμε το τι ζημιά κάνει σε ποια είδη ένα είδος αλίας. Όπως ξέρετε λοιπόν σε διάφορες χώρες ε, που θίγονται έχουν ε, υπάρξει σοβαρές αντιδράσεις, έχει ζητηθεί να επιστραφεί στην Κομισιόν αυτό το έγγραφο και δεν έχει επιχειρηματολογήσει επαρκώς για αυτή την απαγόρευση. Δεν έχουν γίνει σοβαρές επιστημονικές μελέτες για την ε, περιβαλλοντική ε, επίπτωση για τα διάφορα είδη παρασυρωμένων δικτύων, δικτυών όπως εφαρμόζονται, όπως χρησιμοποιούνται σε διάφορα κράτη-μέλη. Γιατί πρέπει να κάνουμε μια σαφή διάκριση μεταξύ των ε, μεγάλων σκαφών που χρησιμοποιούν αυτά τα δίκτυα και τα μικρά σκάφη που χρησιμοποιούν άλλο είδο εξοπλισμού. Δεν έχει να κάνει με τη διαστάσει του ματιού. Έχει να κάνει με, το, με τα μεγάλα σκάφη. Αντίθετα με την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ε, μικρής κλίμακας αλληλεία στην περιοχή μου δεν έχει καμία εναλλακτική λύση. Επαναλαμβάνω, είναι επιλεκτική αυτή η ε, μέθοδος Νομίζω επίσης ότι ε, είναι παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας. Και παραλαμβάνω, δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση αυτής της απαγόρευσης. Δεν είναι λοιπόν αναλογική, αναλογικά κατάλληλη σε σχέση με αυτό που επιδιώκεται. Βεβαίως μπορώ να συμφωνήσω με την πρόταση του συγητή για να απαγορευτούν ορισμένα δίκτυα που βλάπτουν ε, τις, ε, τους θαλάσσιους φυσικούς πόρους. Πρέπει λοιπόν η διαδικασία αυτή να ακολουθήσει η μελέτη αυτή, συγγνώμη, η πρόταση αυτή να βασιστεί σε μια μελέτη να ακολουθηθεί η συνήθις νομοθετική διαδικασία. Δεν είναι δυνατόν να τα αφήσουμε όλα αυτά σε κατ εξοδότηση πράξη της Κομισιόν. Έχουμε χρόνο, πρέπει να αντιμετωπίσουμε ορθά αυτό το θέμα. Συνήθις λοιπόν διαδικασία. Πρώτα απ' όλα μελέτη αντικτύπου για κάθε είδος αλίας που θέλουμε να ε, θίξουμε. Μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ, συνάδελφο Καπούτα από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Με ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αφρόντε για το έργο του συζητητή. Θεωρώ ότι είναι καλή η έκθεσή του αν και νομίζω ότι θα υπάρξουν και κάποιες ε, τροπολογίες. Η σημερινή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα παρασυρώμενα πλάδια παρουσιάζει κάποια κενά. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για τη χρήση αυτών των εργαλείων ε, και ε, ούτε ρυθμίστε δυνατότητα να υπάρχουν στο σκάφος άλλα δίκτυα. Έτσι λοιπόν αυτό επέτρεψε στους Ελλήνες να χρησιμοποιούν τέτοια παρασυρώμενα απλά διαδίκτυα τα οποία απαγορεύονται και αυτό οδηγεί σε πολύ μεγάλους φόβους ό,τι αφορά ε, την ε, διατήρηση των πόρων. Επομένως, θετικά ερμηνεύουμε την πρόθεση της Κομισιόν να παρέμβει για να εγγυηθεί μεγαλύτερη προστασία των προστατευόμενων ειδών όπως είναι οι θαλάσσιες χελώνες, τα κοιτόδη και οι καρχαρίες. Όμως ε, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την απαγόρευση όλων των παρασυρώμενων δικτυών. Επομένω, θεωρούμε ότι είναι δυσανάλογη αυτή η ολική απαγόρευση και θα μπορούσε να έχει κοινωνικό οικονομικό αντίκτυπο πολύ αρνητικό στην βιώσιμη ελεία, στη βιώσιμη ελεία και στι μικρέ κοινότητε. Ο εισηγητή εφιστά την προσοχή μα ορθώ σε αυτά τα σημεία. Νομίζω όμω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια, να βρούμε μια λύση που να καλύπτει όλες αυτές τις πτυχές, δηλαδή και την προστασία των θαλάσσιων ειδών, αλλά και να προστατεύει και αυτόν τον τομέα της αλίας. Εγώ άκουσα κάποιες προτάσεις, μάλλον συγγνώμη έχω κάποιες προτάσεις που θα μπορούσαν να λαμβάνουν υπόψη αυτές τις απαιτήσεις. Θα ήθελα να προτείνω την εισαγωγή του Unnet Rule, δηλαδή να απαγορεύει ε, στους αλείς να έχουν εργαλεία στο σκάφος ε, διαφορετικά δίχτυα μέχρι την 1η Ιουνίου του 2017. Εγώ συμφωνώ με τη βούληση ε, του εισηγητή να απαγορευτεί αυτό το ίδιο του δικτύου που λέγεται φερετάρα. Ε, πρόκειται για ένα δίχτυ το οποίο έχει πάρα πολύ μικρό μάτι, πολύ μικρό μέγεθος ματιών. Νομίζω ότι αν ε, ε, λάβουμε υπόψη το πόσο χρησιμοποιείται το δίκτυο αυτό θα έπρεπε να απαγορευτεί. Έχουμε ένα δίκτυο που έχει πολύ κατώτερο μάτι των 50 ε, χιλιοστών και επομένως ενώ ναι, θεωρώ ότι αν χρησιμοποιηθούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια, χρήση της φερετάρα θα μπορούσε και να επιτραπεί αν λάβουμε υπόψη τον αρνητικό αντίκτυπο αυτού του κοινωνισμού στις παράκτιες κοινότητες, νομίζω πρέπει να προβλέψουμε μια τροπολογία που ε, θα χορηγεί ένα τμήμα του κονδυλίου ένα τμήμα κονδυλίων συγγνώμη, του Ταμείου για τη Θάλασσα σε αυτούς τους αλείς, έτσι ώστε ε, μέχρι τις 31 Μαΐου του 2017 τουλάχιστον να μπορούν να χρησιμοποιούνται αυτά τα εργαλεία. Η θέση μου για αυτή την ε, γνωμοδότηση είναι να προσπαθήσουμε να μετριάσουμε όλες αυτές τις αντιθέσεις και να καλύψουμε όλες τις απαιτήσει. Ευχαριστώ κύριο Ντάνκαν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση αυτή δεν εξυπηρετεί το σκοπό της. Τελεία. Για χρόνια μας λένε ότι η κοινή αλληλευτική πολιτική θα αντιμετωπίσει τα πράγματα σε περιφερειακή βάση. Όμως έτσι δεν είναι τα πράγματα εδώ. Η μικρή αλία στο Ενωμένο Βασίλειο που έχει πιστοποιηθεί από τον αρμόδιο οργανισμό μας λέει ότι αυτή, ε, αυτή η αλία θα καταστραφεί αν εφαρμοστεί αυτό το μέτρο. Έχει χαθεί η αρχική φιλόδοξη ιδέα από την αδέξια προσέγγιση του one size fits all. Δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σαν όλα τα παρασυρώμενα για να είναι ίδια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως πρέπει να δείχνουν τις ίδιες μεταχείρισεις. Για το λόγο αυτό λοιπόν η πολιτική μου ομάδα δεν μπορεί να στηρίξει την πρόταση όσο έχει. Θα πρέπει να παραπεμφθεί εκ νέου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να υπενθυμίσουμε στο όργανο αυτό ότι εφόσον, αρχίζει, ε, εφόσον μιλεί για περιφερειοποίηση να αρχίσει και να την εφαρμόζει, να αναγνωρίσει διαφορές, να προβλέψει διαφορετική μεταχείριση και να μεταχειριστεί με διαφορετικό τρόπο τους αλληλείς που εξαρτώνται από τις αλληλευτικές αυτές μεθόδους. Γιατί αλλιώς βλάπτει σοβαρότατα την εξοπιστία των θεσμικών οργάνων και την δική της την ίδια. Μάλιστα. Η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είπε τίποτα για την γνωμοδότηση ο κύριος Ντάνκαν, μόνο για την αρχική πρόταση επιτροπής. Πρώτα λοιπόν εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα τον εισηγητή που βρίσκεται τα λέει πολύ καλά και που γνωρίζει για ποιο πράγμα μιλεί. Είναι κρίσιμο πραγματικά να συνεχιστεί η μεταρρύθμιση της κοινή ε, πολιτικής αλίας και να προστατεύσουμε τις θάλασσες. Και βέβαια θέλουμε να συνεχιστεί η εκμετάλλευση των θάλασσων και βέβαια θέλουμε να συνεχιστεί η αλία, αλλά θέλουμε να ε, προστατεύσουμε τη βιοπικιλότητα. Και βεβαίω πρέπει να προστατεύσουμε τα προστατευόμενα είδη. Και βέβαια θέλουμε να συνεχιστεί η αλία από την άλλη Σωστό. Γι' αυτό και συμφωνώ απόλυτα με την βασική γραμμή της νομοδότησης του εισηγητού. Ξέρω ότι η άλλη επιτροπή είπε να πάει η πρόταση πίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω επίσης ότι η πρόταση ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι πολύ ευτυχής, α το πω έτσι. Είναι και ευτυχή. διότι μια συνολική απαγόρευση των παρασυρώμενων απλαδιών χωρί βάση δεδομένων, χωρί εξαιρέσει, δεν μπορεί να είναι σωστή. Γιατί έτσι τιμωρεί και εκείνου οι οποίοι χρησιμοποιούν μικρότερα παρασυρώμενα απλάδια και επομένως και την βιοτεχνική εντό εισαγωγικών αλία. Α, από τη Σκοτία δεν είστε εσεί. Ναι, βλέπετε λοιπόν, να, τουλάχιστον στις ακτέ της Ιρλανδίας τα ίδια πράγματα διαπιστώνουμε. Ότι πολλοί χρησιμοποιούν τα δίχτυα αυτά με τρόπο περιορισμένο. Και αυτό είναι σωστό και να συνεχιστεί αυτό. Στην Βαλτική δεν επιτρέπεται καθόλου η χρήση των παρασυρώμενων απλαδιών. Και αλλού και η απαγόρευση του φερετάρας μου φαίνεται σωστή. Πρέπει να δει κανεί βεβαίω ποιε επιπτώσει θα έχει στην αλία, γιατί δεν θέλουμε να απογορεύσουμε την αλία. Μου φαίνεται και η πρόταση των σοσιαλιστών σωστή. Να δούμε εάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ίσω αν μπορούν να ληφθούν χρήματα δηλαδή, από το Ταμείο Αλία για να χρηματοδοτηθούν κάποιε μεταβάσει σε αλίες πιο βιώσιμε. Πάντω γενικά σωστό είναι τα παρασυρώμενα πλάδια των 2,5 χιλιόμετρων που απαγορεύονται ήδη να παραμείνουν υπό απαγόρευση και ειδικότερα στη Μεσόγειο. Κατά τα λοιπά, θεωρώ σωστό και λογικό μου φαίνεται το θέλουν να, να ζητήσουμε τις χώρες μέλη να εξετάσουν πού διεξάγεται μικρή βιώσιμη που θεωρείται ακόμα βιώσιμη, δεν ξέρουμε βεβαίως για πόσο θα μπορεί να θεωρείται βιώσιμη αλία, αυτή να μπορεί να ε, συνεχίσει να εφαρμόζεται. Όμως, οπωσδήποτε να γίνει συλλογή δεδομένων. Κρίσιμο σφάλμα της ε, πρότασης της Επιτροπής, ότι δηλαδή προχωρεί χωρίς επιστημονική βάση. Τα είπε και η συνάδελφός μας του Λαϊκού Κόμματος. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε οπωσδήποτε σε θεμελιωμένη βάση. Αυτά τα, λέει, τα κάνει και η Επιτροπή, αυτά τα λέει και η Επιτροπή Αλίας, ότι πρέπει να βασίζονται σε αυτά τα δεδομένα που έχουν συλλέξει οι επιστήμονες. Νομίζω ότι ανέπτυξα την άποψή μου, ως Επιτροπή Περιβάλλοντος οφείλουμε να προσέχουμε, να τηρούμε την βιοπικιλότητα, να την σεβόμαστε. Η κατεύθυνση είναι σωστή, αλλά χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση. Και γι' αυτό θεωρώ ότι η γνωμοδότηση είναι πράγματι όρθη και την υποστηρίζουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Ροδρίγες. Κατανοούμε ότι πραγματικά βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση ο κλάδος. Έχουμε υπερελίευση που έχει βοηθηθεί από επιδοτήσεις που δόθηκαν στο μεγάλο βιομηχανικό στόλο. Ε, ε, αλία με παρασυρώμενα δίχτυα, ε, θέτει σε κίνδυνο τη θάλασσα και αυτό έχει αποδεικτεί και δυστυχώ υπήρχε συστηματική παραβίαση τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε κάποιε περιοχέ. η έλλειψη εναρμόνισης τη νομοθεσία και η ανεπαρκή ε, έλεγχη επέτρεψαν αυτή η πρακτική να συνεχίζεται με ατιμορρησία κυρίως στη Μεσόγειο η βούληση της απερχόμενης επιτροπής να προωθήσει την εναρμόνιση της νομοθεσίας είναι καλοδεχούμενοι γιατί έχουμε συνεχείς παραβιάσεις σήμερα και διευκολύνονται επειδή υπάρχει ποικιλομορφία νόμων. Παρ' όλα αυτά, ο κανονισμός με την πλήρη απαγόρευση έχει ένα θεμελιώδες πρόβλημα. Το πρώτο είναι ότι δεν αντιμετωπίζει επί της ουσίας το πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, δηλαδή ότι επιστώνουμε την επιτυχία, δεν προχωρά στη δημιουργία μηχανισμών ελέγχου και κυρώσεων για την παράνομη ελεία. Θέλει να είναι ένα κανονισμός με μηδενικό κόστος, όμως αυτό δεν λύνει το πραγματικό πρόβλημα που είναι ο μη σεβασμός της νομοθεσίας. Δεύτερον, η απόλυτη απαγόρευση φοβόμαστε ότι μπορεί να πλήξει την ερασιτεχνική μορφή αλίας που πρέπει να την περισπίσουμε. Παραδείγματο χάρη αναφέρθηκε μια μορφή αλία στην ε, Γαλλικία, έχουμε και άλλες ε, μορφές αλίας που πρέπει να τις υπερασπίσουμε. Πρέπει να υπερασπίσουμε ε, και τα επαγγέλματα, πρέπει να βρούμε μια εναλλακτική στο σημερινό μοντέλο αλίας που αποδεκατίζει τις θάλασσες μας και αυτό θα το κάνουμε με τις βέλτιστες πρακτικές στην παραδοσιακή αλία, στην αλία μικρής κλίμακας. Πρέπει να έχουμε ένα πιο βιώσιμο σύστημα αλίας στο μέλλον. Έτσι λοιπόν, ε, δεν θεωρούμε ότι είναι αποδεκτή η πρόταση της Κομισιόν ούτε ποσοτικά ούτε ποιοτικά μιλώντας από περιοριστική σκοπιά. Χαιρετίζουμε λοιπόν την πρόταση του εισηγητή να αφήσει μια προθεσμία για την εφαρμογή του, κανονισμού της απαγόρευσης και Θέλουμε να προωθήσουμε επιστημονικές μελέτες για την ε, εραστεχνική αλία, να δούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος και να την προστατεύσουμε. Καταλαβαίνουμε ότι ε, αν ε, έχουμε πλήρη απαγόρευση και ανοίξουμε την πόρτα σε διάφορες παρεκκλήσεις που θα εφαρμόζονται ένα κράτος μέλος, θα είναι αντιπαραγωγικό. Εμείς θέλουμε λοιπόν να συνεχίσουμε να το συζητούμε αυτό. Η προηγούμενη εμπειρία μας δείχνει ότι ένα σύστημα παρεκκλήσεων καταλήγει σε μια νομική πολυπλοκότητα και τελικά εξυπηρετεί ακριβώ το αντίθετο από αυτό που επιζητούμε, μια ενερμονισμένη νομοθεσία που να μας διευκολύνει να ελέγξουμε την παράνομη αιλία, η οποία πραγματικά βλάπτει τις θάλασσές μας. Αυτή η νομοθεσία θα έπρεπε να περιλαμβάνει ήδη ρητές προϋποθέσεις για να προστατεύει τα συστήματα της μικρής αιλίας και τα είδη που υπερελέγχουν Γι' αυτό αυτή τη στιγμή οι θέσει μα είναι να αξιολογήσουμε την αναγκαιότητα μια νέα πρόταση κανονισμού που να λαμβάνει κατά νου αυτέ τι δύο αρχέ, τον έλεγχο τη κυρώση, την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και κατά δεύτερον την προστασία και την προώθηση της μικρής παραδοσιακής ελίας που είναι το μοναδικό μέλλον για τη βιώσιμη ελεία στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ο, κύριος Ο Μπάς. Λείπει η σκιώδης μας. Μιλεί αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή Αλίας. Ε, έτσι, επομένω έχει μια σοβαρή δικαιολογία που λείπει. Πολλά λέχθηκαν ήδη. Ευχαριστώ τον εισηγητή που κατέβαλε προσπάθεια να καταλήξουμε σε μια θέση καλύτερη κάπως από το να πούμε απλώς «Α, στείλτε το έγγραφο πίσω στην Κομισιόν». Κάτι που μου φαίνεται υπεραπλουστευτικό. Άκουσα βέβαια και την προσέγγιση του Ιαν Τάνκαν. Αλλά βέβαια η συζήτηση δεν είναι και νέα. Ολόκληρες γενικές συνελεύσεις έχουν ασχοληθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 90 των Ηνωμένων Εθνών εννοώ με ψηφίσματά τους. Ξέρω βέβαια ότι οι Τόριδες έχουν κάποια προβλήματα με τις διεθνείς οργανώσει αλλά μέχρι τώρα δεν πίστευα ότι τους ενοχλεί και η Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ. Έτσι λοιπόν το θέμα δεν είναι νέο, το συζητούμε εδώ και πολύ καιρό. Υπάρχει νομοθεσία από το 1992 και από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι ότι κάθε φορά που συζητούμε την νομοθεσία αντιλαμβανόμαστε βέβαια ότι μια συνολική απαγόρευση δεν μπορεί να λειτουργήσει. Από τη στιγμή όμως που αρχίζουν οι αποκλήσεις ανοίγουν και παραθυράκια. Και άμα ανοίξει παραθυράκια στο νόμο Ανοίγει και τη δυνατότητα καταχρήσεων. Χρειάζεται λοιπόν να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Μπράβο σας λοιπόν εισηγητά που κάνετε την προσπάθεια να ακολουθήσετε αυτόν τον δρόμο που δεν είναι εύκολος. Δεν έχουμε εμείς ε, ακόμη αποκρισταλώσει άποψη ως πολιτική ομάδα. Ευχαρίστως όμως θα συνεργαστούμε με τον εισηγητή και με τις άλλες πολιτικές ομάδες. Συγχαίρω την κυρία Μάισνερ για παράδειγμα για τις απόψεις της αλλά και την ενωτική αριστερά. Νομίζω θα καταλήξουμε σε μια θέση χρήσιμη που να συμβάλλει σε μια πρόθεση της συζήτησης και όχι απλά να πούμε όχι στείλτε το πίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί κάτι τέτοιο ίσως ε, να μην είναι πολύ χρήσιμο. Ερώτηση προς την Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για μια προσφυγή λόγω παραβιάσεως κατά της Ιταλίας. Ακούσαμε ότι αυτή η προσφυγή κατά της Ιταλίας στην περίπτωση αυτή έχει αποσυρθεί δεν ξέρουμε ποιο είναι το περιεχόμενο της υποθέσεως. Μπορείτε να μας πείτε πού βρίσκεστε και εάν όντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποσύρει την προσφυγή. Τότε γιατί. Και αναμένω βέβαια να διεξαχθεί ενδιαφέρουσα συζήτηση για μια πιο χρήσιμη θέση από το να πούμε απλά όχι. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο Μπριάννα που προέρχεται από την Επιτροπή Ελίας και είναι η αρμόδια συγκήτρια για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ελπίζω ότι ε, το γεγονό ότι παρευρίσκομαι εδώ να σας βοηθήσει για να συνεχίσουμε μια σοβαρή συζήτηση σε ένα πολύπλοκο θέμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φρόντε για τη δουλειά που έκανε καθώς και για το πόσο μας βοηθά για τη συζήτηση στην Επιτροπή Ελίας. Εγώ διάβασα εις βάθος ε, την γνωμοδότηση και θεωρώ ότι συνάδει με τη συζήτηση που έχουμε τη δική μας Επιτροπή μεταξύ όλων των ομάδων. Η πρόταση που έκανα ως εισηγήτρια, αν και ακόμα είναι σε ένα στάδιο ακρόασης, ε, γιατί ζητήσαμε και μια επιπλέον ακρόαση της Επιτροπής για τη μελέτη αντικτύπου, και θέλουμε να συζητήσουμε και με τον νέο Επίτροπο. Εμείς είμαστε εντελώς αντίθετοι σε μια πλήρη απαγόρευση έτσι όπως έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως ε, ανησυχούμε και για το γεγονό ότι κάποιοι πρότειναν να απορρίψουμε εντελώς ε, ε, αυτή την νομοθεσία και να την ξαναστείλουμε πίσω στην Κομισιόν. Αντίθετα, εγώ νομίζω ότι έχουμε καθήκον να εργαστούμε επί αυτή τη πρόταση, στη λογική που πρότεινε ο Μαρκοφρόντε, για να προβούμε σε αποσυφήνιση. Γιατί αν διαβάσουμε όσα μας ήρθαν από την Κομισιόν, οι προτάσεις που θα μπορούσαμε να έχουμε ήταν τέσσερις. Η μία ήταν αυτή της διατήρησης του status quo, δηλαδή όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, όμως σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα του ελέγχου, όλοι θεωρήσαμε ότι είναι κάτι αρνητικό. Κατόπιν είχαμε άλλες δύο πιο μεσαίες μετριοπαθείς προτάσεις, δηλαδή να κάνουμε μια αξιολόγηση ανά τρόπο αλίας και ένα ελευτικό εργαλείο και να βρούμε διάφορες λύσεις και η τέταρτη ήταν αυτή που έστειλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τελικά κομισιόν της πλήρους απαγόρευσης. Οι διάμεσες θέσεις όμως είναι οι πιο ενδιαφέρουσες και εγώ προσωπικά και χάρη και στη βοήθεια της Επιτροπής ΕΝΒΗ θα ήθελα να εργαστώ επ' αυτών. Να έχουμε όμως κατά νου ότι για την γνωμοδότηση αφρόντε νομίζω ότι υπάρχουν ε, πολλές ε, θετικές πτυχές. Θα ήθελα όμως να επισημάνω δύο σημεία που πρέπει να αξιολογήσουμε. Δηλαδή να μην προβούμε σε περαιτέρω ε, πολυπλοκότητα, να είναι δυνατόν να υλοποιηθεί η πρόταση αυτή και επίσης να αφήσουμε και μια διακριτική ευχέρεια. Έτσι λοιπόν, ε, αυτά τα δύο θα πρόσεχα και θα ενίσχυε και μία από τις αρχές κλειδιά της κοινή ελευτικής πολιτικής, ε, το θέμα της περιφερειοποίησης. Από τη μελέτη των ελευτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται πριν να μιλήσουμε για διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη Γαλλική και στη Βόρεια Ευρώπη, σύμφωνα με τις ε, διάφορες περιφέρειες όπου χρησιμοποιούνται, θα πρέπει να δούμε και τον αντίκτυπο στο οικοσύστημα, γιατί είναι διαφορετικός. Έτσι, λοιπόν, αυτό θα μπορούσε να είναι μια λύση, είτε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, είτε στην Επιτροπή Ελίας. Εγώ θα ήθελα να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εκπονήσουμε μια νομοθεσία που να επιλύει τα προβλήματα που υπάρχουν αφενός, αλλά και αφετέρου να μας επιτρέψει να προωθήσουμε τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος μαζί με την βιωσιμότητα του ελευτικού κλάδου γιατί πραγματικά έχει πληγεί τα μάλα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Η έκθεσή του προσπαθεί να βελτιώσει την πρόταση της Κομισιόν που είναι απόλυτα μη αναλογική ή κάνει το πιο εύκολο, δηλαδή να απογορεύσει πλήρως τα παρασυρώμενα δίκτυα. Με αυτόν τον τρόπο καταργούμε ένα μεγάλο τμήμα της μικρής κλίμακας ε, αλίας. Θα ήταν καλύτερα να υπάρχει επιλεκτική απαγόρευση για τέτοια δίκτυα που πραγματικά απειλούν. Μιλάω από πλευράς και των συναδέλφων του Μπενεγά και καλό το Κοινοβούλιο να επαναπέμψει την ε, πρόταση στην Κομισιόν διάφορες περιοχές όπως και η Γαλλική από την οποία προέρχομαι έχουν ε, μικρής κλίμακας αλεία που χρησιμοποιούν τα δίκτυα που λέγονται ντεσέιτο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κρεμόμενο ε, από τη μία πλευρά σε ένα μικρό σκάφος λιγότερο από 12 μέτρα και από την άλλη μεριά ε, ε το... Ε, ε, σε μια σημαδούρα. Αυτά τα σκάφη αφορούν ε, ολόκληρες ε, κοινότητες και, και πόλεις όπως, το, όπως η δική μου έχουν 170 τέτοια σκάφη και επιπλέον καταναλώνουν πολύ λίγο ντίζελ. Υπάρχουν λοιπόν έθνη ε, όπως η Γαλλικία που λαμβάνουν υπόψη και τους κανόνες αυτούς για την αλληλεία στα εσωτερικά τους ύδατα που είναι σαν φιόρτ της Ρίας και άρα δεν μπορεί να βασιστεί με βάση την αρχή της επικουρικότητας μια νομοθεσία ε, να εφαρμόζεται σε αυτές τις περιοχές. Από πλευράς του Μπενεγά θεωρώ ότι η κυβέρνηση της Γαλλικίας και της Ισπανίας ε, δεν έκαναν το καθήκον τους, δεν έστειλαν σαφή πληροφόρηση για την κοινωνικο-οικονομική επίπτωση μιας τέτοιας μέτρα, ενός τέτοιου μέτρου στην Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Σουίτσα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Αφρόντε και η άποψή μου συμπίπτει με αυτή τη συναδέλφου Μέισνερ. Είναι πολύ εύκολο να έχουμε μια πλήρη απαγόρευση και είναι πολύ εύκολο να τα αναθέσουμε και όλα στην Κομισιόν. Το δικό μας καθήκον ως μέλη του Κοινοβουλίου είναι να βρούμε μια συμβιβαστική λύση. Συμφωνώ με όσους λένε ότι η κοινή ελευτική πολιτική είναι πράγματι μια περιφερειακή πολιτική. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια περιφερειακή προσέγγιση και τελικά πρόκειται για μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως θα πρέπει να βρούμε μια λύση στη Μεσόγειο έχουμε διάφορα είδη αλευτικών εργαλείων, δικτυών που χρησιμοποιούνται. Ίσως ε, τη δική μου χώρα δεν την ενδιαφέρει τόσο πολύ, αλλά εγώ θα ήθελα να συνεισφέρω την άποψή μου. Αν είχαμε μία ολική απαγόρευση για αυτά τα ελευτικά εργαλεία θα είχαμε αρνητικό αντίκτυπο στην ελευτική δραστηριότητα. Θα πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε και τους μικρούς αλείς και να βρούμε πιθανές λύσεις. Εμείς ως βουλευτές της Επιτροπής Περιβάλλοντος θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα και της προστασίας των οικοσυστημάτων. Επομένως, η μόνη δυνατή λύση είναι συμβιβασμός. Εγώ είμαι υπέρ του να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Και θα ήθελα να προτείνω να συνεχίσουμε την εκπόνηση επιστημονικών μελετών. Γιατί είναι διαφορετικό να συζητούμε από πολιτική σκοπιά χωρίς να υπάρχει επιστημονική βάση. Επίσης, πρέπει να κάνουμε μια διαφοροποίηση μεταξύ των διάφορων αλλιευτικών εργαλείων. Εδώ μιλάμε και διαφορετικά μη δικτυών αλλά και σκαφών. Εγώ λοιπόν είμαι υπέρ ενό διαλόγου γιατί είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο το ζήτημα και νομίζω ότι είναι το καθήκον μας να καταλήξουμε σε μια δυνατή λύση. Ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό. Είχαμε κάποιες ε, ερωτήσεις. Θα δώσω το λόγο στην κυρία από την, στον κύριο Ντονατέλα από την Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή, τον κύριο Αφρόντε, για την επιτελεστή εργασία που έκανε προσπαθώντας να συνοψίσει σε μία έκθεση διάφορες εναλλακτικές λύσεις και τονίζουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για την συζήτηση για το θέμα αυτό μεταξύ των ε, θεσμών. Ευχαριστώ και την κυρία Μπριάνο που είναι συγγήτρια στην Επιτροπή Ελίας και θα έχει δύσκολο καθήκον για να καταλήξει σε μια συνένεση και η προσέγγιση της ε, είναι πολύ θετική. Όλες αυτές οι ροές είναι πολύ σημαντικές για την Κομισιόν. Συζήτηση για το περιεχόμενο της πρότασης που κάνει η Κομισιόν προς, την Επιτροπή, προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Λοιπόν, επί της ουσίας τώρα. Υπενθυμίζω ότι διεξήχθη για πάνω από 1,5 χρόνο μία πολύ αναλυτική μελέτη αντικτύπου για τη χρήση των παρασυρωμένων δικτυών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση αυτή είναι δημοσιευμένη. Για πρώτη φορά υπήρξε τέτοιο επίπεδου μελέτη που έχει δημοσιευθεί και αφορά το είδος και αφορά τη χρήση ενός συγκεκριμένου εξοπλισμού. Είναι κάτι που θα πρέπει να το κάνουμε και σε άλλες περιπτώσεις. Για μας είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό, όχι μόνο για την ε, προετοιμασία προτάσεων, αλλά και για τη δημόσια συζήτηση που πρέπει να διεξάγεται για τα θέματα αυτά. Θα επανέλθω σε αυτό. Έχουμε λοιπόν την μελέτη αντικτύπου. Έχουμε τα επιστημονικά δεδομένα. Ίσως να θεωρείτε ότι δεν υπάρχει επαρκής περιβαλλοντική επίπτωση. Μπορεί να ισχύει αυτό. Αλλά οπωσδήποτε έχουμε ευρεία έκταση ε, τεκμηρίωση για τη χρήση αυτού του είδους δίκτυων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούστηκε επίσης ότι δημιουργούν πρόβλημα ορισμένες προτάσεις για το εύρος εφαρμογής της πρότασης, ότι αφορά τα πάντα. Ότι δεν έχει υπάρξει επαρκής περιφερειακή διαφοροποίηση, που είναι μία αρχή της νέας ε, κοινή ελευτικής πολιτικής. Νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο, ίσως όχι σήμερα. Η περιφερειοποίηση σημαίνει ότι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα που έχουν κάποιες περιφέρειες. Εμείς όμως ξέρουμε ότι η χρήση αυτού του εξοπλισμού στο εσωτερικό των κρατών μελών και σε διάφορα κράτη-μέλη δεν μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε την αρχή της περιθυροποίησης. Δηλαδή, δηλαδή, Ό,τι αποφασί και αν λάβουμε πρέπει να αφορά την αντιμετώπιση του κινδύνου αλίευσης ε, απειλωμένων ή απειλουμένων ή προστατευομένων ειδών. Ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές όχι μόνο της Μεσογείου αλλά και του Ευξήνου και του Ατλαντικού. Θέλουμε λοιπόν μια πρόταση που να αντιμετωπίσει αυτόν τον κίνδυνο. Χρειάζεται να είμαστε πιο επιλεκτικοί να εξετάσουμε κάποιες ιδιαιτερότητες. Βεβαίως, να το κοιτάξουμε μαζί με το Κοινοβούλιο. Και με βάση την έκθεση που υποβάλλατε σήμερα υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Όπου υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουμε προσέγγιση. Βεβαίως, να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση με βάση το έγγραφο που θα διατυπώσετε και εδώ εσείς ε, ως ένβη αλλά και στην ΠΕΣ. E Κάτι άλλο για τα στοιχεία. Από τη στιγμή υποβολής της πρότασης έχουμε λάβει μεγάλης έκτασης ε, συμπληρωματική πληροφόρηση από τα κράτη-μέλη, από εμπλεκόμενους φορείς, από το πώς διεξάγεται αυτή η αλληλεία στην Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε την πρωτοβουλία να ξαναγράψει το Σεπτέμβριο στα κράτη-μέλη για να εξασφαλίσει επιβεβαίωση κάποιων στοιχείων που μας είχαν αποσταλεί ορισμένες φορές άτυπα. Τώρα λαμβάνουμε αυτές τις επιβεβαιώσεις. Είναι σαφές ότι λείπουν κάποια στοιχεία από την αρχική μελέτη αντικτύπου. Γιατί κάποια στοιχεία για κάποιο λόγο δεν απεστάλησαν στην Κομισιόν έγκαιρα. Τα είχαν τα κράτη-μέλη, δεν θεώρησαν ότι είναι αρκετά σημαντικά, δύσκολο να πούμε, αλλά το σημαντικό είναι ότι ανακαλύπτουμε όλο και περισσότερες ε, τέτοιου τύπου δραστηριότητες κάθε μέρα. Ανακαλύπτουμε λοιπόν όλο και περισσότερα στοιχεία που θα βοηθήσουν να διευκρινίσουμε το πλαίσιο για τη διαχείριση της χρήσης παρασυρωμένων. Και όπως κάναμε και για τη μελέτη αντικτύπου, Φυσικά τα στοιχεία αυτά να σας τα αποστείλουμε. Τα στοιχεία που λαμβάνουμε από τα κράτη-μέλη καθημερινά, για να έχουμε όλοι την ίδια τεκμηρίωση για τη δραστηριότητα αυτή, την επίπτωσή τους και τους κινδύνους που ενέχει. Ελπίζω λοιπόν ότι σύντομα θα έχουμε όλα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να συμπληρώσουμε την αρχική μελέτη αντικτύπου. Και τέλος, τέλος, για να απαντήσω μια ερώτηση για την προσφυγή κατά της Ιταλίας. Το 1992 είχαμε ήδη απόφαση του δικαστηρίου, διότι δεν υπήρχαν σωστές διαδικασίες ελέγχου και επίβλεψης από τις Ιταλικές αρχές και κάποια θέματα αφορούσαν την ε, ασάφεια της Ιταλικής νομοθεσίας που, επέτρεπαν, που επέτρεπε αυτή η ασάφεια στους αλληλείς να χρησιμοποιούν απαγορευμένα τέτοια δίκτυα. Αυτά λέει η απόφαση του 1992. και η Ιταλία δεσμεύτηκε να εφαρμόσει ένα πολύ εκτεταμένο πρόγραμμα δράσης και αυτή τη δέσμευση την ανέλαβε το 2011. Το πρόγραμμα αυτό δράσης είναι ένα επίσημο έγγραφο που εγκρίθηκε και από το Σώμα των Επιτρόπων και το πρόγραμμα δράσης εφαρμόζεται και επιτηρείται η εφαρμογή του και από τις Ιταλικές Αρχές και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ως αποτέλεσμα της εφαρμογής, οι πολιτικές ελέγχου της Ιταλίας έχει πλήρως αναδιαμορφωθεί και βελτιωθεί. Οι μεγάλες κλίμακες παράνομες ε, δραστηριότητες τέτοιας αλίας με βάση την πληροφόρηση που έχουμε και την πληροφόρηση που έχει συλλέξει η Ιταλία, η τέτοιου τύπου λοιπόν αλία είτε έχει πλήρως σταματήσει ή είναι πλέον πολύ χαμηλού επίπεδου και τέτοιου τύπου χαμηλού επίπεδου παράνομες δραστηριότητες ε, γενικά παρατηρούνται. Δεσμεύθηκε λοιπόν η ειναι πλεον πολυ χαμηλου επιπεδου και τετοιου τυπου χαμηλου επιπεδου παρανομες δραστηριοτητες γενικα παρατηρουνται δεσμευτηκε λοιπον η ιταλια και γι' αυτό η Κομισιόν έκλεισε την υπόθεση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παρακολουθούμε την εφαρμογή. Σημαίνει ότι όσον αφορά αυτήν την δικαστική απόφαση αποφασίσαμε ότι δεν χρειάζεται να συνεχιστεί η εφαρμογή. Συνεχίζουμε όμως να παρακολουθούμε την κατάσταση ούτω ώστε στη Μεσόγειο να ε, υπάρχει μόνο νόμιμη αλήθεια. Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Αφρόντα για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Πολλά θα είχα να πω, αλλά δεν θέλω τώρα να καθυστερήσουμε. έχει χρόνο, γιατί θα αναβάλουμε το επόμενο σημείο. Έπρεπε να φύγει ο συνάδελφος Νταντέν. <laughs> Θα ήταν καλύτερα να μου το είχατε πει μάλλον. Εντάξει, εντάξει, με τριοπαθώς να χρησιμοποιήσετε το χρόνο. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι αρκετά πολύπλοκος αυτός ο φάκελος, επομένως μια τέτοια συζήτηση γίνεται πολύ χρήσιμη γιατί μας δίνει πάρα πολλά στοιχεία προς προβληματισμό. Και πρέπει να πω ότι χάρηκα πολύ που είδα, που η δουλειά που έκανα, που δεν ήταν και απλή, σας διαβεβαιώ, εκτιμήθηκε. Γι' αυτό δράτω την ευκαιρία να ευχαριστήσω ειλικρινά τη γραμματεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος που έκανε μια τεράστια δουλειά για να μεταφράσει τις ιδέες μου σε ένα έγγραφο το οποίο να μπορεί να είναι παρουσιάσιμο. Πολύ καλή δουλειά της γραμματείας. Λοιπόν, ορισμένα σημεία για τα όσα υπόθηκαν, ορισμένα σχόλια για τα όσα υπόθηκαν. Φυσικά θα αναφερθώ σε όλους όσους μίλησαν και θα αξιολογήσω τόσο υπόθηκαν και θα τα αποτιμήσω. Κάποια συγκεκριμένα σημεία. συνάδελφος Καπούτα έδωσε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες και μπορώ να πω ότι θα τις υποδεχτώ θετικά στη διαδικασία των τροπολογιών, δηλαδή η απαγόρευση το να υπάρχουν επί το σκάφος διάφορα εργαλεία είναι κάτι πολύ σημαντικό, μου διέφυγε και ευχαριστώ που μου το επιθυμήσατε. Επίσης και ταμείου για να βοηθήσουμε τους ε, αλλοί σε αυτό το μεταβατικό στάδιο είναι κάτι εκτιμητέο. Είμαι πάντοτε πολύ προσεκτικός όταν μιλάμε για κονδύλια, γιατί πάντοτε έχει υπάρξει κατάχρηση στον τομέα της ελίας των κονδυλίων, αλλά αν μιλάμε εδώ για λύσεις που θα πρέπει να προβούν σε αναπροσαρμογή, σίγουρα καλό να τους βοηθήσουμε κατά κάποιο τρόπο. Πολλοί συνάδελφοι υπογράμμισαν πόσο σημαντικό είναι να εργαζόμαστε με επιστημονικά δεδομένα στις περιπτώσεις αυτές. Στοιχεία που να είναι και ποιοτικά και ποσοτικά καλά. Η πρότασή μου προς αυτήν την κατεύθυνση πηγαίνει. Δεδομένου ότι προφανώς υπήρξε πρόβλημα στη συλλογή των δεδομένων και ο ίδιος εκπρόσωπος της Κομισιόν μόλις μας είπε ότι τώρα φτάνουν τα στοιχεία και εμείς εργαζόμαστε επί μιας πρώτης Κομισιόν που έχει παρουσιαστεί όμως. Προφανώς λοιπόν έλειπαν κατά τη σύνταξη της πρότασης αυτής τα στοιχεία. Έτσι λοιπόν, εγώ σκέφτομαι να ακολουθήσω αυτή την κατεύθυνση και να πω ότι σε αυτή την ε, περίοδο παρέκκλησης ε, θα τη χρησιμοποιήσουμε για να συλλέξουμε σημαντικά στατιστικά στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να απαγορεύσουμε με ακρίβεια μόνο τα εργαλεία τα οποία έχουν πολύ μεγάλη επίπτωση στο περιβάλλον. Για να απαντήσω τώρα σε ορισμένους συναδέλφους που είπαν ότι θα προτιμούσαν ε, να ξαναστείλουμε πίσω το φάκελο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι όπως είναι. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με τη θέση αυτή. Εμείς τώρα έχουμε την μπάλα στο γήπεδο μας ως ε, κοινοβούλιο, πρέπει να τοποθετηθούμε, να πούμε την απόψή μας και από τη στιγμή που ασκούμε κριτική στη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το καθήκον μας είναι να πούμε ποιες είναι εναλλακτικέ και τι θέλουμε εμείς να προκύψει από τη συζήτηση αυτή. Να ξαναστείλουμε πίσω το φάκελο λοιπόν, θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ εύκολο και πλουστευτικό. Εδώ εμείς είμαστε για να εργαστούμε και να βρούμε λύσεις. Κάτι άλλο που άκουσα. Ξέρω ότι η διαδρομή που αναφέρω στην γνωμοδότησή μου είναι πολύπλοκη. Ξέρω ότι ε, να δώσουμε την ευθύνη ακόμη και για μια συγκεκριμένη περίοδο και κατά παρέκκληση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα γιατί εσύ δίνεις την ευθύνη, αναθέτεις την ευθύνη σε ένα, στατό, σε ένα κράτος μέλος χρησιμοποιώντας την παρέκκληση είναι πάρα πολύ εύκολο να ε, βρεθούν εκεί ε, κάποια κενά στην νομοθεσία. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια επικίνδυνη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να φοβόμαστε αν ε, εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι θέλουμε να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα, να αποκτήσουμε μια πραγματική προστασία του περιβάλλοντος και αυτό θέλουμε να το κάνουμε μέσω της συλλογή δεδομένων και της ενημέρωσης των κρατών μελών, ε, είναι ένα κίνητος που πρέπει να αναλάβουμε, αν η πρόταση που έχω κάνει φυσικά χρήζει και βελτίωσης, αλλά αν η πρόταση που έχω κάνει θετηθεί, νομίζω ότι ε, μπορούμε να τη συζητήσουμε, να επιφέρουμε κάποιες νέες ιδέες και προτάσεις και τελικά να καταλήξουμε στο εξή και να πούμε ότι ως Επιτροπή Περιβάλλοντος έχουμε καταλήξει στο αποτέλεσμα το δικό μας που είναι το εξή. Να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την προστασία του περιβάλλοντος και για τα προστατευόμενα είδη που πλήττονται από αυτά τα δίκτυα χωρίς ε, να είναι δυνατόν να υπάρχει πολύ μεγάλος αντίκτυπος ε, στις μικρές ελευτικές κοινότητες. Και αναφέρθηκαν πάρα πολλέ φορέ σήμερα το πρωί, χρησιμοποιούν κάποια δίκτυα που δεν έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον, αλλά και στηρίζουν και την οικονομία τους με αυτή την αλία. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Περιμένω τις τροπολογίες σας. Και πραγματικά με καθησύχασε η συζήτηση αυτή. Θεωρώ ότι έχουμε ακολουθήσει τη σωστή κατεύθυνση και εύχομαι να έχουμε καλό αποτέλεσμα γιατί κατόπιν ε, θα πρέπει να πάμε και να συζητήσουμε και με τη συνάδελφο στην Επιτροπή Ελίας. Δεν θα είναι εύκολο ούτε εκεί. Είναι και εκεί η συζήτηση πάρα πολύ έντονη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα εγώ να υπενθυμίσω το χρονοδιάγραμμα, προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών και θα προτιμούσα να έχουμε ψηφική βεβαίωση 10 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 3 Δεκεμβρίου τον Ιανουάριο θα ψηφίσει η Επιτροπή Αλίας και θα πάμε στην Ολομέλεια στις 2 Φεβρουαρίου. Και τώρα να σας πω ότι θα αναβάλουμε το σημείο 18 για την επόμενη συνεδρία της Επιτροπής μας, γιατί ο συνάδελφος Νταντέν ε, έχει αποχωρήσει. Θα το δούμε λοιπόν στην έκτατη συνεδρία της Επιτροπής μας και ε, Δευτέρα στο Στρασβούργο. Σας ευχαριστώ λοιπόν και μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ολοκληρώσαμε τη συνεδρίασή μας.